ότι συνιστά την πρώτη οδηγία στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης που προσδιορίζει κοινού κανόνες για μετανάστες χαμηλής ειδίκευσης. Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης. Όπως γνωρίζετε, η επεξεργασία του σχεδίου οδηγίας για την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών με στόχο την ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση ξεκίνησε το 2010. Πρόκειται για σημαντικό νομοθετικό εργαλείο. Η οδηγία αυτή αναμένεται αφενός να δημιουργήσει το κοινό πλαίσιο κανόνων για μια νέα ταχεία διαδικασία εισόδου και διαμονής για τους ενδοεπιχειρησιακά μετακινούμενους και αφετέρου να οικοδομήσει έναν μηχανισμό απλών και σύντομων διαδικασιών κινητικότητας των υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα της κινητικότητας συνιστά τη μείζωνα προστιθέμενη αξία της εν λόγω οδηγίας. Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης οδηγίας μπορεί και πρέπει να ολοκληρωθεί στους αμέσως επόμενους δύο ή τρεις μήνες και οπωσδήποτε εντός αυτής της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλά έχουν μέχρι σήμερα επιτευχθεί ως προς τούτο. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για τις επίμονες και επίπονες προσπάθειές τους τόσο τον εισηγητή της Επιτροπής, της Επιτροπής τον κύριο Γιακολίνο, όσο και την εισηγήτρια της Επιτροπής Απασχόλησης, Κυρία Γιάκουσας, ζητούμε από πλευρά σας να επιδείξετε ευελιξία στις προσπάθειες της ελληνικής προεδρίας. Πρέπει να συγκεράσουμε το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ευέλικτη διαδικασία κινητικότητας με τους προβληματισμούς των κρατών μελών τόσο για τη διασύνδεση του συστήματος με το Σέγγεν όσο και για την αποφυγή καταχρήσεων και κακής εφαρμογής των ρυθμίσεων της ε, οδηγίας. Θα πρέπει να επιτευχθεί η συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου εντός της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου επί των εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν κυρίως στην ίση μεταχείριση, στη διατήρηση ημί παράλληλων ευνοϊκότερων συστημάτων εισδοχής και στον υποσυζήτηση μηχανισμό κινητικότητας. Καλούμε και την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιδείξει αντίστοιχη βούληση και πρόθεση προς την κατεύθυνση αμοιβαίων παραχωρήσεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας άμεσα δεδομένων και των ασφικτικών προθεσμιών. Εμείς ως Προεδρία σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση λαμβάνοντας υπόψη και τις ευαισθησίες που έχετε προς τούτο επιδείξει. Πρόταση οδηγίας αναδιατύπωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εισδοχή και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας, των σπουδών, της ανταλλαγής μαθητών, της αμοιβόμενη και μη εκπαίδευσης του εθελοντισμού και της εσωτερικής άμυστης βοήθειας. Όπως γνωρίζετε η πρόταση οδηγίας για την αναδιατύπωση των οδηγιών για τις σπουδέ και τους ερευνητές, η επεξεργασία της οποίας ξεκίνησε πρόσφατα, στοχεύει στα παρακάτω. Πρώτον, να καταστούν τα εφιστάμενα νομοθετικά εργαλεία πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά. Δεύτερον, να μετατραπούν οι δυνητικές διατάξεις της οδηγίας για τους σπουδαστές, τους εθελοντές και τους άμυστους ασκούμενους σε υποχρεωτικές και τρίτον να εισαχθούν δύο νέες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών, οι έμιστοι ασκούμενοι και οι εσωτερική άμυστοι βοηθή περισσότερο γνωστή ως ΟΠΕΡ. Η πρόταση οδηγίας έχει τύχει επεξεργασίας στο πλαίσιο των αρμοδίων ομάδων εργασίας του Συμβουλίου κατά το τελευταίο οκτάμινο ενώ παράλληλα η Επιτροπή σας έχει προχωρήσει αρκετά επί του σχεδίου οδηγίας. Δεδομένων των ασφικτικών περιορισμών από την περάτωση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο στόχος της ελληνικής προεδρίας εστιάζεται στην μεγαλύτερη κατά το δυνατόν προώθηση των σχετικών συζητήσεων. Η βούληση της ελληνικής πλευράς θα ήταν η προώθηση των συζητήσεων με στόχο την έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας με το σημερινό Συμβούλιο. Επ' αυτού υπάρχουν δύο προβλήματα. Αφενός η πρόταση οδηγίας για τους ενδοεπιχειρησιακά μετακινούμενους είναι πολύ πιο όρημη και πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί. Αφετέρου τα σημεία που χωρίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη δείχνουν να είναι ακόμα αρκετά στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερο την εισηγήτριά σας επί της πρώτας οδηγίας, αγαπητή κυρία Σεσίλια Βίξτριμ, καθώς χάρη στις επίπονες προσπάθειές της έχουμε ήδη αναχείρας τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από πλευρά σας είναι σημαντικές και μας δίδουν σε κάποιες περιπτώσεις λύσεις σε προβλήματα που έχουν ανακύψει στο πλαίσιο των ομάδων του Συμβουλίου. Πάντως θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση η Προεδρία θα επιδιώξει ό,τι καλύτερο μπορεί υπό τις δεδομένες συνθήκες αλλά και τα ασφικτικά πλέον χρονικά περιθώρια. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάσαμε τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας για το επόμενο εξάμεινο. Γνωρίζουμε ότι οι προκλήσεις και οι δυσκολίες είναι πολλές. Ευελπιστούμε ότι κατά το εξάμεινο της ελληνικής προεδρίας θα οθήσουμε με ουσιαστικό τρόπο τα πράγματα με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του χώρου της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας στην Ένωση. Είμαι στη διάθεσή σας για όποιες ερωτήσεις θέλετε να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ κύριε κύριε Μιχελάκη, κύριε Υπουργέ Εσωτερικών, για την εισήγησή σας. Ανακοίνωσα ότι θα έπρεπε να ακούσουμε καταρχήν τις τρεις εισηγήσει και μετά να έχουμε ένα γύρο ερωταπαντήσεων από τους ευρωβουλευτές, ξεκινώντας με τους συντονιστές. Αλλά μόλις μου είπαν ότι ο κύριος Αθανασίου, υπουργό Δικαιοσύνης, θα μας εγκαταλείψει για να πάει σε κάποια άλλη συνεδρία στις 4 και 4. Τώρα όμως είναι ήδη 4 ε, παρά τέταρτο. Οπότε ίσως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τώρα ένα πρώτο γύρο ερωταπαντήσεων, εάν ε, συμφωνείτε κύριε Γενική Γραμματέα, εάν συμφωνείτε κι εσείς, έτσι ώστε να μπορέσει να μπορέσουμε να ακούσουμε πρώτα τις ερωτήσεις που απευθύνονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης και να μπορέσει και εκείνος ε, να απαντήσει με τη σειρά του. Ε, να ξεκινήσουμε λοιπόν με τους συντονιστές, γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε το χρόνο. Τι έχετε να πείτε, διαδικαστικό κύριε Κάσον? Όχι, απλά σηκώνετε το χέρι για να υποβάλλετε ερώτηση, μάλιστα. Ωραία λοιπόν, ξεκινάμε με τους συντονιστές. Κυρία Ματία, Ματιέ, με συγχωρείτε, εσείς πρώτοι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Ελληνική Προεδρία και τους υπουργούς που μας έκαναν ε, εξονυχιστικές εισηγήσεις και για το ότι είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Ε, κύριε Υπουργή, είναι μια προεδρία που φαίνεται να είναι εξ αρχής κάπως περίπλοκη γιατί είναι το τέλος της θητείας και είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση για κάθε φορά για την προεδρία. Είναι πολύ φορτωμένες νομοθετικά περίοδοι και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχηθώ καλό κουράγιο για αυτή την ε, προεδρία. Κύριε Αθανασίου, μιλήσατε για διάφορα θέματα και προτεραιότητες πολύ πολύ ενδιαφέρουσες. Εγώ ήθελα να σας θέσω κάποιες ερωτήσεις, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο μαζί σας. Καταρχήν, μιλήσατε για το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του Ρέζης, ε, πολύ σημαντικά θέματα. Ε, μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι πολύ σημαντική για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, καταρχήν ξέρετε ποια είναι η πρόταση της Κομισιόν, βρίσκεται επιτάπητος, ενώ έχουν ε, διάφορα κράτη-μέλη βγάλει κίτρινη κάρτα για όλα αυτά και θα ήθελα να γνωρίζω αν και όσον με αφορά εγώ είμαι απόλυτα υπέρ της δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μάλιστα θα ήθελα να επεκταθεί και το πεδίο εφαρμογής αλλά δεν έγινε αυτό δυνατό μέχρι στιγμής. Θα ήθελα να ξέρω εσείς Προς τα πού θα οθήσετε αυτό το θέμα. Φαντάζεστε μια ενισχυμένη συνεργασία έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το θέμα εάν κάποια κράτη-μέλη εξακολουθήσουν να είναι επιφυλακτικά για αυτό το θέμα. Και έπειτα μιλήσατε για την ενιαία θηρίδα. Ε, μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω και έπειτα για το θέμα της προστασίας των δεδομένων, data protection. Προς ποια κατεύθυνση θα πιέσετε έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες καθώς να μπορούν να ε, συμφωνήσουν και εκείνοι για αυτό το θέμα που είναι πολύ σημαντικό για αυτή τη θητεία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μωράης. Εάν κατάλαβα καλά κύριε Πρόεδρε, θέλετε να υποβάλουμε ερωτήσεις μόνο προς τον Υπουργό Αθανασίου για την ώρα. Καταρχήν να ευχηθώ στην Ευρωπαϊκή Προεδρία και σε εσά κύριε Υπουργέ καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Εσείς είστε υπεύθυνο για το πακέτο της προστασίας των δεδομένων που είναι μεγάλη προτεραιότητα της Προεδρίας. Σας ευχαριστώ πολύ επίσης που αναφέρατε την έρευνα για την μαζική παρακολούθηση που θεωρούμε ότι είναι ένα κομμάτι του συνολικού πακέτου που θα θέλαμε να δούμε ως τμήμα ε, του κανονισμού και της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο αισιόδοξο είστε όσον αφορά μια ψηφοφορία τον Μάρτιο και για το ότι δεν θα μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο σε σχέση με κάποια πιο δύσκολα σημεία του εις δέσμης. Δεν μπορούν να επιτευχθούν πολλά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και μάλιστα σε μια προεδρία που διακόπτεται από τις ευρωεκλογέ. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πόσο αισιόδοξο είστε. Και έχω και άλλες ερωτήσεις για τους άλλους δύο υπουργού, αλλά αυτή τη στιγμή ήθελα μόνο να θέσω την ερώτηση από τη δική μου ομάδα για το θέμα του πακέτου συνάδελφος θα σας ρωτήσει για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Φαντάζομαι ότι θα θέσει αυτή την ερώτηση γιατί είναι σκιώδης υπεύθυνη για αυτό το θέμα. Αλλά έτσι και αλλιώς και το ΕΛΚΑ έθεσε αυτή την ερώτηση. Thank you, Chair, and thank you to the ministers for their uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τις εκτεταμένες σας εισηγήσεις. Έχω διάφορες ερωτήσεις και δεν είμαι βέβαιος ότι τις απευθύνω προς το σωστό Υπουργό γιατί σχετίζονται περισσότερο με θέματα που δεν ανεφέρθησαν και δεν ξέρω σε ποιο το χαρτοφυλάκιο εμπίπτουν. Το ένα θέμα που ανεφέρθη είναι η NSA και όλες αυτές οι μαζικές ε, παρακολουθήσεις και τα σχετικά σκάνδαλα. Είμαι ευτυχής που αναφέρθηκε γιατί μέχρι στιγμής ε, στην ουσία ε, μια ηχηρή σιωπή μόνο έχουμε ακούσει από το Συμβούλιο. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν αν συζητιέται το θέμα στο Συμβούλιο πέρα από τις συζητήσεις το, κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών γευμάτων που δεν κρατώνται πρακτικά. Έπειτα, οι απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Ομπάμα θεωρείται ότι είναι αρκετές και έπειτα το Συμβούλιο θα υποβάλει δικές του προτάσεις. Και κάποια άλλα θέματα που δεν ανεφέρθησαν, το ένα είναι η μεταρρύθμιση του κανονισμού περί διαφάνειας, η πρόσβαση στα έγγραφα, για τα οποία ο κύριος Κάσμαν που είναι εδώ παρόν είναι συγητής μας. Πιστεύω πως όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, μια πολύ άσχημη κατάσταση όσον αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Πιστεύω πως είναι σκανδαλώδες οι Κομισιόν και το Συμβούλιο να αρνούνται να προχωρήσουν και να καταστήσουν πιο διαφανή και όχι λιγότερο διαφανή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο εγώ σίγουρα δεν μπορώ να εξηγήσω στους ψηφοφόρους μου τον Μάιο. Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω πού βρισκόμαστε σε αυτήν την αποκαλούμενη οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων που κάπως έχει εξαφανιστεί, μια μαύρη τρύπα την έχει ρουφήξει από ό,τι φαίνεται. Είναι κάτι το οποίο είναι προς όφελος των πολιτών και έπειτα υπάρχουν και διάφορα άλλα θέματα τα οποία εμπίπτουν πάνω κάτω στην εντολή της Επιτροπής μας και που δεν είναι απαραίτητο θέματα προεδρίας, αλλά είναι θέματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Και επειδή θα έχετε την Προεδρία, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσετε κι εσείς στην χώρα σας αυτά τα προβλήματα. Θα ήθελα να ξέρω πώς βλέπετε την κατάσταση, όπως για παράδειγμα καταπολέμηση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής. ποιε είναι οι απόψεις σας όσον αφορά την ελευθεροτυπία, τον πλουραλισμό, την αντιμετώπιση των ετούντων άσυλο και τέλος της αυξανόμενη ρατσιστικής βίας κατά των ε, των φιλομεταβατικών ε, που από ό,τι ξέρω υπάρχουν σχετικές έρευνες από πλευράς της αστυνομίας. Μάλιστα, ο κύριος Χρυσόγελος από πλευράς των Πρασίνων. Έχετε το λόγο. Ε, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργή, καλώς ήρθατε. Είναι μια δύσκολη προεδρία και έχετε να διαχειριστεί πολύ σημαντικά θέματα, όπως για παράδειγμα αυτό που είπαν και προηγούμενοι συνάδελφοι, το θέμα της μαζικής παρακολούθησης πολιτών και επιχειρήσεων από την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας των ΗΠΑ. Ε, περιμένουμε από τη δικιά σας Προεδρία τουλάχιστον να μας ενημερώσετε ποια μέτρα πρόκειται να πάρετε, ιδιαίτερα όταν διεξάγονται παράλληλα και οι συζητήσει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για τις εμπορικές σχέσεις. Το Κοινοβούλιο είχε ασκήσει πολύ έντονη κριτική και για τη συνέχιση αυτών των σχέσεων. Ε, περιμένουμε τουλάχιστον από το ε, από την ελληνική προεδρία να μας ενημερώσει αν υπάρχει κάποια πρόοδο στα θέματα αυτά. Ε, το δεύτερο είναι ότι ξέρουμε ότι σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα υπάρχει μια αυξανόμενη παρουσία ακροδεξιών και ρατσιστικών οργανώσεων και το θέμα της Χρυσή Αυγή ξέρετε ότι είναι και, δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα αλλά αφορά συνολικά όλη την Ευρώπη. Για πολύ καιρό όμως τα ρατσιστικά εγκλήματα ήταν ατιμόρυτα. Ξέρετε ότι στον Ισαγγελέα πήραν πολλές υποθέσεις που δεν είχαν διαρευνηθεί. Ε, υπάρχει μια αιτιολόγηση γιατί τέτοια εγκλήματα δεν είχαν ε, εξεταστεί στο παρελθόν και έπρεπε να φτάσουμε στη δολοφονία κάποιου Έλληνα για να ξεκινήσει η δικασία και για άλλους που κυρίως ήταν μετανάστες. Ε, και ποια είναι η πρόοδος των ερευνών σε σχέση με το χαρακτηρισμό της χρυσή αυγή ως εγκληματικής οργάνωσης ε, ή και ως οργάνωση προετοιμάζονταν για ανατροπή του, ε, του, της δημοκρατίας, δημοκρατικού πολιτεύματος. Τα Επίσης υπάρχουν τα θέματα των ε, διακρίσεων, όπως αναφέρθηκαν και προηγούμενοι συνάδελφοι, και κατά πόσο η ελληνική προεδρία δεσμεύεται τώρα να εφαρμόσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το σύμφωνο συμβίωσης και την άρση όλων των διακρίσεων που φορούν άτομα LGBT κλπ. Ξέρω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι δυνατόν η ελληνική Προεδρία να μην εφαρμόζει αυτά που ζητάμε να εφαρμοστούν από τα Δυτικά Βαλκάνια ή από τρίτε χώρες και περιμένουμε στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας να εφαρμόσετε αυτό που όλη η Ευρώπη υποστηρίζει και όλα τα πολιτικά κόμματα υποστηρίζουν. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι εξαίρεση. Και τέλος τα θέματα του ξεπλήματος ε, χρήματος και της διαφοράς. πολλές περιπτώσεις όπως είναι μίζες στη διάρκεια εξοπλιστικών προγραμμάτων έχουν περάσει μέσα από offshore εταιρείε όπου εμπλέκονται και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις π.χ. γερμανικές επιχειρήσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων και περιμένουμε η Ελληνική Προεδρία να δείξει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στα θέματα της αντιμετώπισης διαφθοράς και να ακολουθήσει και κάποια στοιχεία από τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση διαφθοράς. Περιμένουμε να δούμε κάποιες πρωτοβουλίες από την Ελληνική Προεδρία ε, πάνω στους τομείς. Okay, Mr. for the... Ο κύριος Κέρκοπ για τους συντηρητικούς. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο, Τρία σημεία έχω. Καταρχάς, θα ήθελα να ρωτήσω πώς ε, σκοπεύει η Ελληνική Προεδρία να αντιμετωπίσει τα σοβαρά και συνεχιζόμενα θέματα ασφαλείας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα για τους Ευρωπαίους πολίτες που φεύγουν από την Ένωση και ριζοσπαστικοποιούνται τους ξένους μαχητές, ξένους στρατιώτες. Δεν ήθελα να μου πείτε την απόψή σας. Έπειτα, σκοπεύει η Προεδρία να θέσει ως προτεραιότητα την ε, συζήτηση που έχουμε εδώ για την ε, ανάγκη μιας ε, συμφωνίας για τα δεδομένα των επιβατών με τρίτες χώρες μέχρι την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Και τρίτον, η ελληνική προεδρία έχει θέσει ως προτεραιότητα το άσυλο και τη μετανάστευση για το εξάμεινό της. Είναι ενθαρρυντικό, ε, ενθαρρυντική αυτή η στήριξη που βλέπουμε για μεγαλύτερη ετοιμότητα στην ε, Μεσόγειο. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν ε, σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το χρονικό διάστημα και για να δημιουργήσετε τη δική σας μακροπρόθεσμη προσέγγιση σχετικά με τους τούτες άσυλο και τους πρόσφυγες στα κέντρα κράτησης στην Ελλάδα και στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Τριανταφυλίδης για την ΚΟΕ excuse Η κυρία Βερζιάτ πρώτα, με συγχωρείτε. Ε, αντικαθιστώ το συντονιστή μας, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη γι' αυτό. Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύσκολη για τη χώρα που την αναλαμβάνει, ειδικά όταν υπάρχει και προεκλογική περίοδος παράλληλα. Το να έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι να λάβει ευθύνε ευθύνες και σίγουρα η χώρα σου μπαίνει στο προσκήνιο και χύνεται το φως στα τεκτενόμενα της χώρας Προεδρίας. Κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, κύριε Θεμασίν, τελειώσατε την πανέβασή σας λέγοντας ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν θα υποστούν κανένα περιορισμό και τον εξασφαλίσουμε το κράτος δικαίου είναι πολύ σημαντικό. Κανένας δεν είναι κάτω από τον νόμο ή υπεράνω του νόμου και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτή την άποψη. Όμω. <clears throat> Διάφορε συνδικαλιστικέ οργανώσει και ΜΚΟ, καθώ και οργανώσει ε, υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μα επέσαν την προσοχή για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Η κατάσταση είναι αρκετά ανησυχητική. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην υγεία αμφισβητούνται από αυστηρές περικοπές ε, στις δημόσιες ε, δαπάνες, λόγω της λιτότητας. Έχουμε λοιπόν ε, φαινόμενα βίας, φαινόμενα καταπίεσης ε, λόγω αυτού. Καταγγέλλονται τέτοια φαινόμενα. Η Ελλάδα έχει ευθύνη σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Γιατί είναι ο βασικός, ε, η βασική πύλη εισόδου αυτών των μεταναστών. Αυτά, αυτοί οι μετανάστες όμως είναι και θύματα βίας. Αμφιζητώνται τα πιο θεμελιώδη δικαιώματά τους. Ε, υφίσταται κακή μεταχείριση. Αυτό το καταγγέλουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η αστυνομία ακόμα μερικές φορές εμπλέκεται και είναι υπέτεια. Η Ελλάδα καταδικάστηκε μάλιστα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ακριβώς για τέτοια θέματα. Διάφοροι συναδελφοί μου μίλησαν για ρατσισμό. Χρειάστηκε να γίνει η δολοφονία του Παύλου Φίσα για να κινητοποιηθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Βεβαίω δεν είναι μόνο η Ελλάδα εκεί υπεύθυνοι. Αλλά στην Ελλάδα σε 17% των υποθέσεων αυτών εμπλέκεται και η αστυνομία και η αστυνομία έχει ύποπτο ρόλο. Ε, μιλήσαμε πολύ για το κλείσιμο της ΕΡΤ και ορισμένοι ε, δημοσιογράφοι μάλιστα αντιμετωπίζουν και ποινικέ δίκες. Όλα αυτά μας ανησυχούν πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι φυσικό να μας δώσετε κάποιες συγκεκριμένες, στοχευμένες απαντήσεις για αυτά τα στοιχεία. Ε, και για αυτέ τι καταγγελίες των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Μιλάμε για μη κυβερνητικέ οργανώσει με τι οποίες ε, δουλεύουμε χρόνια. Ε, παραλληλίζουν την Ελλάδα με την Ουγγαρία και θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, να μας απαντήσετε εάν πρόκειται να σας πιστέψουμε, κύριε Υπουργέ, για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και κάτι πιο συγκεκριμένο τώρα. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κείμενο για τη διάσωση στη θάλασσα. Θα ήθελα να μάθω τη θέση της ελληνικής προεδρίας για αυτό το κείμενο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Thank you all. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τώρα το γύρο των ερωτήσεων από τους συντονιστές. Είναι τέσσερις ακριβώς. Ο Υπουργός κ. Αθανασίου θα πρέπει να φύγει, όπως σας είπα, στις 4 και τέταρτο. Προτείνω λοιπόν τώρα να έχουμε τον πρώτο γύρο απαντήσεων από τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Μιχελάκη και μετά θα προχωρήσουμε με τις ερωτήσεις των υπόλοιπων μελών αφού ακούσουμε τον Γενικό Γραμματέα κύριο Γεωργιάδη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις. Είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρουσες και θα χρειάζονται Εμπεριστατωμένη απάντηση. Θα ήμουν ευτυχής αν είχα περισσότερο χρόνο να απαντήσω πιο διεξοδικά και σε άλλες ερωτήσεις, αλλά θα προσπαθήσω μαζεύοντας τις ερωτήσεις σε ενότητες, σε ενότητες να μπορέσω να είμαι όσο μπορώ πιο ε, σαφής και να απαντήσω σε όλες. Λοιπόν, για τα προσωπικά δεδομένα. Η Ελληνική Προεδρία θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειες της επί του φακέλου της προστασίας των δεδομένων. Έχουμε προγραμματίσει πολλές συναντήσεις για το σκοπό αυτό. Είναι πάνω από 20, τουλάχιστον 20 συναντήσεις θα έχουμε. Σε τεχνικό επίπεδο. Θα προχωρήσουμε τις εργασίες επί της οδηγίας και όπως ε, ανέφερα και στην ε, εισήγησή μου, όπως έκανε η Ιδανική, η Κυπριακή, η Ιρλανδική και η Λιθωνική Προεδρία, θα υποφεληθούμε κατά περίπτωση των εργασιών επί του κανονισμού για να προωθήσουμε την πρόοδο των εργασιών. Το θέμα των παρακολουθήσεων από τις υπηρεσίες που αναφέρατε αναφυσβήτητα είναι ένα ζήτημα με υψηλό πολιτικό ενδιαφέρον. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Η ανησυχία του Ευρωπαίου πολίτη που ζει και δρά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έντονη όταν τα προσωπικά του δεδομένα διαβιβάζονται προς τρίτες χώρες. Η κοινή γνώμη και ο πολιτικός κόσμος έχουν ευαισθητοποιηθεί ακόμη περισσότερο ως προς το ζήτημα αυτό. Το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων όταν αυτά διαβιβάζονται προς τρίτες χώρες πρέπει να είναι επαρκές, ικανοποιητικό, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη ως προς τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Άρα λοιπόν η Ελληνική Προεδρία έθεσε το θέμα αυτό προς συζήτηση στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης που συγκαλείται στην Αθήνα μεθαύριο και θα συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά το θέμα τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Η ενιαία θηρίδα είναι ένα ζήτημα πράγματι που συνεπάγεται ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου όμως χρήζει περαιτέρω συζήτηση ε, στο Συμβούλιο. Θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης Εσωτερικών Επιθέσεων το Οκτωβρίο. Τώρα και την υπόθεση πρίσμου που ετέθη. Η Προεδρία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα προγράμματα παρακολούθησης των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αντίκτυπο στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών. Γνωρίζετε πολύ καλά όλοι τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους διάφορους οργανισμούς η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ εξέτασε τις μαζικές πρακτικές, τις πρακτικές παρακολούθησης. Το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή έχουν μαζί με τις Ηνωμένε Πολιτείες συστήσει μια ατχό κομμάδα ομάδα εργασίας ε, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτή η ομάδα έχει ως έργο να εξετάσει το νομικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες παρακολούθησης των ΗΠΑ που έχουν αντίκτυπο στα προσωπικά, στα πρόσωπα, έχουν αντίκτυπο στα πρόσωπα που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος της ΑΤΧΟ κομμάδος εργασίας έχει ήδη εκδώσει την αναφορά του ε, νομίζω νομίζω τις 27 Νοεμβρίου. Η Επιτροπή επίσης εξέδωσε τον περασμένο Νοέμβριο ανακοίνωση για την επανάκτηση της εμπιστοσύνης στη ροή των δεδομένων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα συζητήσει την αναφορά της ως πιο πάνω εξεταστικής επιτροπής της ΛΥΜΠΕ και προτίθεται να τη συζητήσει το Συμβούλιο. Έχουμε ανησυχίες και θέλω αυτό να γίνει κατανοητό από όλου. Υπάρχουν ανησυχίε και συμμεριζόμαστε και τι ανησυχίε σα. Γι' αυτό τον Απρίλιο, στο Συμβούλιο, στη συνάντηση των αξιωματούχων που θα γίνει με, ε, ε, στην, στην Αθήνα, με αξιωματούχους και των ε, Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχιστεί ο διάλογος για την βελτίωση αυτής της κατάστασης. Τώρα, όσον αφορά τον... Ε, να δω αν έχω κάτι ακόμα για τα προσωπικά δεδομένα. Όχι, να πάμε στον ε, εισαγγελέα. Λοιπόν, Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εγγελικής Αρχής, όπως σας είπα προηγουμένως, θα βοηθήσει στην ε, πάταξη της απάτης σε βάρος των συμφερών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν δυσκολίες για την, ε, ε, για την ψήφιση. Γιατί το λέω αυτό, διότι υπάρχουν συνταγματικές διαφορές στα διάφορα κράτη. Υπάρχει δηλαδή διαφορετική από χώρα σε χώρα συνταγματική ανεξαρτησία. Ας πούμε στη χώρα μας, στην Ελλάδα, υπάρχει μια ζηλευτή δικαστική ανεξαρτησία που δεν παρεμβαίνει καθόλου η εκτελεστική εξουσία. Είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν πάρα ε, πολύ επισταμένος. σα λέω παραδείγματο χάρη ποια θα είναι η δομή τη εισαγγελική αρχή, ποιε θα είναι οι αρμοδιότητες τη, τι σχέση θα έχει ο εισαγγελέα με τι εθνικέ εισαγγελικέ δομέ και τι εξουσίες τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελική αρχή. Η ίδρυση λοιπόν δεν πρόκειται να θίξει, θα προσπαθήσουμε δηλαδή, να μην μπορεί να θίξει τον σκληρό πυρήνα των εθνικών αρμοδιοτήτων της εισαγγελικής αρχής κάθε κράτους μέλους. Αλλά αντιθέτως πρόκειται να ενδυναμώσει και να συσφίξει την περαιτέρω συνεργασία των εθνικών εισαγγελικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή για να έχουμε μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του κοινού σκοπού της ολοκληρωμένης προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της, ε, της Ένωσης. Τώρα, το θέμα της, ε, αν θα πάμε σε μια ενισχυμένη ε, συνεργασία για αυτά, είναι κάτι που θα το δούμε με την εξέλιξη των εργασιών. Είναι κάτι που, δεν αποκλείεται. Θα, και ε, εξάλλου είναι κάτι που προβλέπεται και από την ε, νομοθεσία. Πάντως ε, η τοποθέτηση είναι αυτή ότι αν θέλουμε να έχουμε μια αποτελεσματική αντιμετώπιση της απάτης σε βάρος των συμφερόντων η εισαγγελική αρχή θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή διότι και θα, θα συντονίζει κυρίως θα συντονίζει το έργο των εισαγγελικών αρχών και των κρατών μελών και βεβαίως θα ενδεχομένως ενδεχόμενες παραλήψεις να μπορεί να τις ε, ε, διορθώνει ε, δίνοντας τις απαραίτητες κατευθύνσεις χωρίς βεβαίως να θίγεται όπως σας είπα η ανεξαρτησία των επιμέρους εισαγγελικών αρχών. Ένα ζήτημα που ετέθη για τα δημόσια έγγραφα πρέπει να πω ότι είναι αυτό είναι ένα, δηλαδή για την απλούστευση της αποδοχής των δημοσίων εγγράφων είναι ένα ιδιαίτερα τεχνικό θέμα αυτό και χρειάζεται κάποιος χρόνος για να διαμορφώσουμε τις τελικές θέσεις. Εξαρτάται από, το πρόεδρο, από την πρόοδο των εργασιών στα κατώτερα όργανα. Τώρα, δεν θα μιλήσω για τα θέματα της τρομοκρατίας ε, και τις, ε, το, το θέμα των ξένων μαχητών είναι, θα σας τα πει ο κύριος Γεωργιάδης, είναι της αρμοδιότητός του, να μην χάσω και χρόνο και να ε, πω λίγο για, για τα θέματα τα οποία θίξατε και κυρίως είναι, αφορούν και την χώρα μου. Λοιπόν, έχει υπάρχει μια ε, παρεξήγηση για τη χώρα και επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες οι οποίες είχαν, ε, καθιέρωσαν ε, νόμο για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας από το 1979. Είναι ο νόμος 927 του 1979. Ε, ήταν για την εποχή το ένας νόμος πλήρης αντιμετώπιζε όλο, όλο το φάσμα της ξενοφοβίας και του ρατσισμού βεβαίως σήμερα έχουν αλλάξει συνθήκες και χρειαζόταν μια ε, επικαιροποίησή του και εναρμόνιση με την απόφαση πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη έχει καταρτιστεί νομοσχέδιο, έχει περάσει από την, Επιτροπή, από την αρμόδια Επιτροπή Επεξεργασίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου και σε λίγες μέρες, πολύ σύντομα, θα ψηφιστεί από την ε, Ολομέλεια. Μάλιστα έχουμε προχωρήσει και πέραν από τις ομάδες προστασίας που προβλέπει η απόφαση πλαίσιο και ε, προστατεύουμε και άλλες ομάδες που δεν προβλέπονται στην, ε, στην απόφαση πλαίσιο, όπως παραδείγματο χάρη ε, το θέμα των, ε, των γενετήσεων καταβολών, της αλλαγής φύλου και βεβαίως το, της αναπηρίας. Είναι ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται. Θέλω να σας πω ότι και το συνδυάζω αυτό τώρα με το θέμα που ετέθη με τη Χρυσή Αυγή Πρέπει να ξέρετε ότι ο ελληνικός λαός έχει υποστεί πολλά από τον ναζισμό και τον φασισμό και έχει μεγάλες ευαισθησίες. Τα ποσοστά που βλέπετε της χρυσή αυγή δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες ε, διάκενται και επικροτούν τις αρχές και το πρόγραμμα της χρυσή αυγή. Αντίθετα, είναι ένας ε, λαός καθαρά δημοκρατικός που απεχθάνεται τον ολοκληρωτισμό και τον ναζισμό. Τι γίνεται όμως σε αυτή την περίπτωση. Έχει ε, η οικονομική συγκυρία και πρέπει να το πούμε με θάρρος αυτό και η οικονομική ανέχεια η οποία ήταν ως αποτέλεσμα της αυτής της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας οδήγησε πολλούς ε, πολίτες θα ψηφίζουν ακραία κόμματα. Ένα από αυτό λοιπόν ήταν και η, η Χρυσή Αυγή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Έλλην, οι ψηφοφόροι τους είναι οργανωμένοι στην, ε, στην ε, στη Χρυσή Αυγή. Ε, θα ήθελα να τονίσω εδώ τώρα για την πορεία των ανακρίσεων. Ε, Καταρχή, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όπως ανεφέρθηκα ήδη η ελληνική δικαιοσύνη είναι παντελώ ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία. Ούτε ο Υπουργό Δικαιοσύνη μπορεί να παρέμβει στο έργο τη. Οι ανακρίσει προχωρούν με ταχύ ρυθμό. Ε, έχουν πολλά ηγετικά στελέχη της χρυσή αυγή μετά την απολογία τους έχουν οδηγηθεί στη φυλακή ως ε, προσωρινός κρατούμενο, κρίθηκαν δηλαδή προφυλακιστέοι, αλλά εάν αποτελεί εγκληματική οργάνωση ως σύνολο η Χρυσή Αυγή η προσέξτε τη διαφορά που θέλω να τονίσω, άλλο να πούμε ότι η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση, αυτή καθ' αυτή, και άλλο ότι μέσα στη Χρυσή Αυγή δρούσε εγκληματική οργάνωση. Είναι κάτι το οποίο, για το οποίο θα αποφανθεί η δικαιοσύνη και δεν ήταν ε, σωστό και σόφρον εκ μέρους μου να προδικάσω τις αποφάσεις ε, των δικαστηρίων. Για τους, ε, θα είμαι όμως ειλικρινής μαζί σας. Πράγματι υπόθηκε ότι κατά το παρελθόν πολλές περιπτώσεις ε, βιοπραγίας κατά ξένων και ειδικά μεταναστών δεν ε, οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Ξέρετε γιατί γινόταν αυτό. Γιατί θα σας τα πει βεβαίως και ο κύριος Μιχελάκης ότι το ένα δέκατο του πληθυσμού μας αυτή τη στιγμή είναι μετανάστες. Παράνομοι μετανάστες και νόμιμοι μετανάστες πολλοί από αυτούς δεν κατήγγελαν τις πράξεις βίας. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είχαν, ε, φοβόταν, φοβόταν την απέλαση. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ούτε θέλουμε να κρυφτούμε από αυτό. Πράγματι υπήρξαν περιπτώσεις, ε, περιπτώσεων βίας κατά μεταναστών, οι οποίοι δεν κατήγγελαν τις πράξεις αυτές μόνο και μόνο γιατί φοβόταν την απέλαση. Ήδη όμως ενθαρρύνομαι σήμερα με, μια, με πρωτοπόρα νομοθετικά μέτρα που έχει έχουμε λάβει στην Ελλάδα ε, προστασίας των μαρτύρων και προστασίας των θυμάτων από αυτές τις ε, περιπτώσεις και έτσι έχουμε ε, το τελευταίο καιρό αθρώες καταγγελίες. Υπήρξαν πράγματι ένας συνάδελφος που ανέφερε ότι υπήρξαν ε, μερικές καταδίκες και αστυνομικών. Ναι, υπήρξαν καταδίκες αστυνομικών, δεν είναι αμετάκλητες οι αποφάσεις, θα δούμε, αλλά, υπήρξαν, αλλά είναι εντελώς μεμονωμένες και θα παρακολούσα αυτό να μην γίνει κανόνας ότι ε, η ελληνική αστυνομία δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι δύο-τρεις εξαιρέσεις, οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και αυτοί τιμωρήθηκαν. Τώρα για το θέμα της, ε, της συμβίωσης. Εδώ και πολλά χρόνια από το 2004 ή 2005 ε, στην Ελλάδα καθιερώθηκε και το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ετεροφύλων. Ξέρουμε την απόφαση του δικαστηρίου γιατί καταδικάστηκε η χώρα μας για την ε, ε, απαγόρευση της ότι δεν ενέκρινε δηλαδή την συμβίωση των σε ομόφυλα άτομα. Είναι ένα θέμα το οποίο το εξετάζουμε και θα δούμε σε επίπεδο αστικού οικογενειακού δικαίου ε, είναι και πολιτική απόφαση των κομμάτων της κυβέρνηση και του ελληνικού κοινοβουλίου. Είναι ένα θέμα ανοιχτό το οποίο το εξετάζουμε, δεν έχουμε πάρει απόφαση. Όμως όσοι στρέφονται σε ποινικό δίκαιο, τώρα σε ποινική διαδικασία κατά των ζευγαριών αυτών τιμωρούνται και θα τιμωρούνται αυστηρά από την ελληνική νομοθεσία. Τέλος, για τις, ε, την παιδεία που είπατε. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν, έχουμε πρόσβαση, δεν έχουν πρόσβαση οι ξένοι στην παιδεία και στην ε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σας πληροφορώ ότι ακόμα και οι παράνομοι μετανάστες έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην παιδεία και, και τα παιδιά του, τα παιδιά τους δηλαδή, και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους έχουν ε, πρόσβαση στην αεροτροφορμακευτική ε, περίθαλψη. Και μάλιστα μέχρι πρώτη χωρίς να χρηματοδοτούμεθα ούτε με ένα ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα καταβάλλεται μια προσπάθεια και νομίζω θα υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης για αυτές τις ε, περιπτώσεις. Δεν ξέρω κύριε Πρόεδρε αν παρέλειψα κάτι. Νομίζω ότι κάλυψα το θέμα. Α, το θέμα για τη ε, για τα, τα θαλάσσια σύνορα κλπ. Είναι αρμοδιότητα κυρίως του Υπουργού Εμπορικής Αυτιλίας. Δεν ξέρω όμως αν θα συμπληρώσει κάτι ο κύριος Γεωργιάδης ενώ του ότι τα, τα σύνορα μας όπως ξέρετε είναι εκτεταμένα τα θαλάσσια και πολλοί μετανάστες εισέρχονται από το θαλάσσιο χώρο. Ευχαριστώ πολύ. Okay, as we're coming close to... Μάλιστα, επειδή πλησιάζουμε στις 4 και 4 όπου εσείς θα αναχωρήσετε, είδα να σηκώνονται πάλι χέρια. Έχετε κάποια επερώτηση σύντομα πριν να φύγει ο Υπουργό και μετά θα περάσουμε πρώτα στον ε, Υπουργό Εσωτερικών και μετά θα ακούσουμε και τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ο υπουργό ε, μου είπε ότι πρέπει να φύγει στις 4 και 4. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να ακούσουμε και να... τις απαντήσεις του είναι αυτός. Έχετε κάποια επερώτηση σύντομα, πολύ σύντομα κατάλαβα καλά ότι το Συμβούλιο δεν θα συζητήσει τον αντίκτυπο του σκάνδαλου μαζικών παρακολουθήσεων. Βασικά αυτό είπατε, ότι υπάρχει αυτή η ομάδα εργασίας ε, υπαλλήλων και αυτά. Δεν θα δοθεί καν απάντηση στη δήλωση του Ομπάμα. Σωστά σας κατάλαβα, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει επιτροπή, αναμένουμε το πόρισμα, νομίζω υπάρχει επιτροπή του Συμβουλίου και αναμένουμε το πόρισμα για να το εξετάσουμε. Δεν νομίζω ότι δεν εξετάζεται. Ίσα ίσα έχει μεγάλη ευαισθησία και ο Πρόεδρος και τα μέλη της, ε, ε, της Επιτροπής, οποίοι εξετάζουν με μεγάλη προσοχή και ευαισθησία το ζήτημα αυτό. Okay, Τώρα, κύριε Μιχελάκη, εσείς τώρα θα απαντήσετε και μετά θα περάσουμε στου υπολείπου. Ναι, σα έχω δει όλου. Σα έχω καταγράψει. Όλοι θέλετε να υποβάλλετε ερωτήσει. Παρακαλώ, κύριε Μιχελάκη. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να συμπληρώσω πάνω στο θέμα των ε, δικαιωμάτων των ε, νόμιμων και παράνομων ε, μεταναστών στο θέμα της υγείας και της παιδείας που ακούστηκε και θα ήθελα να δώσω εδώ κάποια στοιχεία. Θέλω να τονίσω εδώ ότι νόμιμοι και παράνομοι μετανάστες έχουν δικαιώματα. Τα παιδιά τους έχουν πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση και στον υπηαγωγείο και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. ξαναλέω, νόμιμη και παράνομη. Πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στις όλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και νηπιαγωγείο. Όσον αφορά το θέμα της υγείας, και αναφέρομαι πάλι στους νόμιμους και παράνομους, ως προς τα παιδιά πλήρη δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες υγείας στα δημόσια νοσοκομεία. Για τους ενήλικες παράνομους έχουμε, έχουν πρόσβαση σε δωρεάν περίθαλψη, σε έκτακτα περιστατικά, σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Όσον αφορά το θέμα του αριθμού των μεταναστών, θέλω να σας δώσω απλώς κάποια στοιχεία για να καταλάβετε σε σχέση με το μέγεθος και τον πληθυσμό της χώρας την ένταση του φαινομένου. Είμαστε 11 εκατομμύρια, είναι 11 εκατομμύρια ο πληθυσμός της Ελλάδος και θα σας δώσω δύο νούμερα για να καταλάβετε το μέγεθος και την πίεση που υφίσταται η Ελλάδα από, την, ε, από τις μεταναστευτικές ροές. Έχουμε λοιπόν 540.000 νόμιμους μετανάστες. 730.000 παράνομους μετανάστες που έχουν, ο αριθμός αυτός προκύπτει από τις συλλήψεις που έχει κάνει η αστυνομία και το λιμενικό σώμα μετά το 2007. Δεν ισχυρίζομαι ότι αυτός είναι ο ακριβής ο αριθμός και οι παράνομοι μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα. Είναι όμως ενδεικτικός ο αριθμός για να καταλάβετε ξαναλέω την πίεση που υφίσταται μια χώρα 11 εκατομμυρίων όσον αφορά την μεταναστευτική πίεση. Μέχρι το 2012 το 90% των παράνομων μεταναστών προς την Ευρώπη έμπαιναν από την Ελλάδα. Εκεί λοιπόν έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ήδη από τα χερσαία σύνορα, την περιοχή του Εύρου, από τότε που φτιάχτηκε το γνωστό τείχος, σχεδόν, τον τελευταίο χρόνο, σχεδόν έχει μηδενιστεί. Το πρόβλημα υπάρχει, αν θέλετε αυτή τη στιγμή, και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, στα θαλάσσια σύνορα όπου γνωρίζετε ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά νησιά. Θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα, στο θέμα της ελευθεροτυπίας που ακούστηκε από κάποιον συνάδελφο. Επιτρέψτε μου εδώ να έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα, καθώς από το 1979 έως το 2011 που ενεπλάκην στην πολιτική εργάζομαι ως επαγγελματίας δημοσιογράφος στον ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, τηλεοπτικούς σταθμούς, ραδιοφωνικούς, εφημερίδες. Πραγματικά, σας λέω, πρόβλημα ελευθεροτυπία στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς, θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω ότι όποιος παρακολουθεί λίγο πιο στενά τα θέματα της ελληνικής επικαιρότητα θα έχει διαπιστώσει ότι ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινής επικαιρότητα έχει να κάνει με τα αποτελέσματα των ερευνών των διοκτικών αρχών και των δικαστικών αρχών όσον αφορά φαινόμενα μαύρου χρήματος, μίζες και οποιασδήποτε φαινομένου διαφθοράς επιχειρηματίες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια αυτή τη στιγμή βρίσκονται προφυλακισμένοι και αν θέλετε όσοι εμπλέκονται είτε αυτοί έχουν σχέση με τον κρατικό μηχανισμό είτε με τον ιδιωτικό τομέα είτε και είναι εμπλεκόμενοι ή είναι προφυλακισμένοι ή διεξάγονται έρευνες πάνω σε αυτές. Και αν θέλετε το μέγεθος της καταπολέμησης διαφθοράς που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι πάρα πολύ μεγάλο για να μπορέσουμε να κλείσουμε με το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα τώρα να πάω σε ένα τελευταίο θέμα <clears throat> στο οποίο έχει τεθεί, διότι εν πολλής ο συνάδελφός μου ο κύριος Αθανασίου κάλυψε τα υπόλοιπα αναφορικά με το θέμα της χρυσή αυγή. Πραγματικά εδώ θα ήθελα να πω ότι οι Έλληνες επειδή έχουν όπως σας είπε και ο κύριος Αθανασίου υποστεί μεγάλα ε, τεράστια, έχει, ματώσει η χώρα από, το, από τους Ναζί και από τους φασίστες, θέλω να σας πω ότι οι Έλληνες ούτε Ναζί είναι, ούτε φασίστες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, ένα κομμάτι της κοινωνίας που λόγω των οικονομικών προβλημάτων, αν θέλετε, κατευθύνεται σε αυτή την ακραία πολιτική οργάνωση. Έχουν να κάνουν με καθαρά οικονομικά θέματα. Δεν είμαστε ούτε ναζί, ούτε ξενοφοβικοί. Οι Έλληνες μετά τον πόλεμο γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας πήγε ως μετανάστες σε πολλές ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες για να εργαστούν. Νομίζω ότι υπάρχουν ελάχιστα σπίτια τα οποία να μην έχουν βιώσει στην οικογένειά τους τη μετανάστευση. Αυτή, ε, αυτός ο λαός δεν είναι ούτε ξενοφοβικός ούτε ρατσιστές. Είναι μια μικρή ομάδα που εκμεταλλεύεται το θυμό και την οργή για τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν. Και πιστέψτε με, η καλύτερη αντιμετώπιση για την εξαφάνιση αυτού του φαινομένου, του φαινομένου της χρυσή αυγή είναι η ανάπτυξη. Και αν θέλετε, η προσπάθεια της χώρας μου είναι να κατευθυνθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, χωρίς να κάνω κατάχρηση του χρόνου, να σας δώσω κάποια οικονομικά στοιχεία, γιατί καλά αυτά που λέω για τις προσπάθειες ανάπτυξης, θα ρωτήσει κάποιος και τι έχετε κάνει πάνω στο σημείο αυτό. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ορισμένα νούμερα. Μέσα σε τέσσερα χρόνια η χώρα μου μείωσε το έλλειμμα κατά 13% του σημερινού ΑΕΠ. Για να το κάνει όμως αυτό, υπέστη μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 25 φορές, κατά 25%. Τη μεγαλύτερη θα ήθελα να τονίσω εδώ, προσέξτε το, μείωση ακαθάριστου εθνικού προϊόντος που έχει υπάρξει ποτέ διεθνώς από τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30. Σε έξι συνεχόμενα χρόνια ύφεσης, ο μέσος Έλληνας έχει χάσει το 38% περίπου του βιωτικού του επίπεδου σε σύγκριση με το 2007. Η ανεργία από το 7% που ήταν σε αυτή τη χώρα έφτασε στο 27%. Για τους νέους δε κάτω των 25 αγγίζει το 60%. Και εύχομαι αυτό το δράμα να μην το περάσει καμία χώρα. Στη διεθνή κατάταξη του ΩΣΑ, η Ελλάδα κατατάσσεται ήδη στην πρώτη θέση διεθνώς στην εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών. Και τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας που έχουν γίνει με αιματηρές θυσίες, με αιματηρές θυσίες ξανατονίζω του ελληνικού λαού, φαίνεται σε όλες τις έρευνες. Ήδη έχουμε ανακτήσει όλη τη χαμένη ανταγωνιστικότητα από το 2002 και μηδενίσαμε το έλλειμμα στο εμπορικό μας ισοζύγιο. Το 2013 για πρώτη φορά η Ελλάδα έβγαλε πρωτογενές πλεόνασμα στα δημοσιονομικά της. Και για πρώτη φορά έβγαλε πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Ενώ για το 2014 φαίνεται, υπάρχουν ήδη όλες οι ενδείξεις, ότι για πρώτη φορά θα σταματήσουμε την κατηφόρα και θα έρθει η ανάκαμψη μετά από έξι χρόνια οδυνηρής και αιματηρής ύφεση. Ζητάω συγγνώμη αν σας κούρασα με αυτά τα νούμερα, όμως αυτή δεν είναι απλή αριθμή. Είναι οι αριθμοί που πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται οι αιματηρές θυσίες ενός λαού. Και αυτό, ξαναλέω για να έρθω στην αφορμή που μου δώσατε για να τα πω και να σας ευχαριστήσω πολύ γι' αυτό ότι αυτή είναι η καλύτερη αντιμετώπιση των ρατσιστικών, ξενοφοβικών, ναζιστικών φαινομένων. Και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Τώρα, όσον αφορά για τις έρευνες που υπόθηκαν, ρώτησε κάποιο συνάδελφος, έπρεπε να υπάρξει μια δολοφονία ενός νέου Έλληνα για να αρχίσουν. Όχι βέβαια. Η οργάνωση αυτή βρισκόταν υπό παρακολούθηση εδώ και αρκετό καιρό. Αν θέλετε, τα στοιχεία που ήρθαν από την τραγική δολοφονία του νέου ανθρώπου, του νέου Έλληνα και τα στοιχεία που είχαν ε, συγκεντρωθεί από τις άλλες έρευνες που είχαν γίνει ήταν αυτές που όπως σας είπε και ο κύριος Αθανασίου οδήγησαν τον αρχηγό της χρυσή Αυγής και στελέχη αυτού του κόμματος να είναι σήμερα προφυλακισμένοι και να περιμένουν την ετιμιγορία του νόμου. Εάν δεν είχαν γίνει έρευνες πριν, ίσως δεν θα μπορούσαμε να έχουμε στοιχειοθετήσει κατηγορίες. Άρα, οι έρευνες υπήρχαν και με αφορμή αυτή την δολοφονία, αυτή την τραγική δολοφονία του Παύλου Φίσα, μαζί με όλα τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, και με τις επιθέσεις σε μετανάστες μπορέσαμε να φτιάξουμε το κατηγορητήριο, να το συγκεντρώσουμε όλο σε ένα φάκελο για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα. Ευχαριστώ. We thank you. We thank you for your... Σας ευχαριστούμε για τις εξηγήσεις σας. Το πάθος με το οποίο απαντήσατε ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ζητώ την κατανόηση τώρα για την, το πρόβλημα που δημιουργείται στην ομαλή διεξαγωγή της ε, συνεδρίασης και στην ε, φάση των ερωτήσεων και απαντήσεων, γιατί τώρα θα ήθελα να απαντήσει ο Γενικός Γραμματέας, ούτως ώστε να μπορέσει και αυτό σε συνέχεια να απαντήσει ερωτήσεις. είναι απαραίτητο να μα κάνει και εκείνο την ομιλία του. Εν συνεχεία θα έχουμε αρκετό χρόνο, ούτω ώστε να δώσουμε σε όλου του ευρωβουλευτέ το λόγο που επιθυμούν για να κάνουν ερωτήσει στους υπουργού, του υπουργού που είναι ακόμα εδώ, δηλαδή ο κύριος Μιχελάκη και ο κύριος Γεωργιάδης. Παρακαλώ, μπορείτε να, ακούσετε, να κάνετε τώρα την παρουσίασή σα. Σα ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ε, οφείλω να απολογηθώ εκ μέρου του Υπουργού Δημοσιαστάξης ε, και Προστασίας του Πολίτη της Ελλάδας, του κυρίου Δένδια, ε, διότι εχθές το βράδυ προέκυψε ε, σοβαρό υπηρεσιακό ε, θέμα και έτσι αναγκάστηκε να αναβάλει την επίσκεψή του με αποτέλεσμα να είμαι εγώ σήμερα μαζί σας. Κατά συνέπεια θα προσπαθήσω κατά το δυνατόν να ανταποκριθώ όσο καλύτερα μπορώ στις απαιτήσεις της ε, Επιτροπή σας. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, καταρχήν οφείλω να σας πω ότι η Ελληνική Προεδρία θα συνεχίσει το έργο της ε, Ιρλανδικής και Λιθουανικής Προεδρίας στο πλαίσιο του προγράμματος του τρίο των Προεδριών και εισαγωγικά θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την επίτευξη συμφωνίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων και με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τους εισηγητές του, τον κύριο Γκυγιόμ, ε, Φοντάνα, Γιακολίνο και Μαρινέσκου για την επικοδομητική προσέγγιση ε, στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Ε, θα ήθελα επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελληνική Προεδρία θα φροντίσει ώστε και οι τέσσερις κανονισμοί που σχετίζονται με το πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους από τους νομικούς γλωσσολόγους θα τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατό. Τώρα, ε, σε σχέση με τον τομέα της παράνομης μετανάστευσης και του ασύλου, ε, είναι γεγονός ότι η επισφαλής ατμόσφαιρα στο εγγύς περιβάλλον της Ευρώπης σε συνδυασμό με την ε, διατηρησιμότητα των γενεσιουργών αιτίων που προκαλούν τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση επιδρούν επαυξητικά στην πίεση που ασκείται στα κράτη-μέλη. Όλα αυτά σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης όταν όλες οι δυνάμεις και οι ενέργειες θα έπρεπε να είναι προσιλωμένες στις μεταρρυθμίσεις για τη διαφύλαξη της σταθερότητας και την αναζωογόνηση της ανάπτυξης. Το βάρος αυτής της πίεσης πέφτει της πίεσης των μεταναστευτικών, των παράνομων μεταναστευτικών ροών, πέφτει όπως είναι φυσικό στα κράτη-μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αυτά τα οποία μαστίζονται από βαθιά ύφεση και υψηλή ανεργία την ίδια στιγμή. Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει την εφαρμογή του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα για την ενίσχυση της αλληλεγγύης στα κράτη-μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου υφίστανται ιδιαίτερη πίεση σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ένωσης και τους διεθνείς οργανισμούς. Ο σεβασμός και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ετούντων ασύλου και των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας θα είναι στην κορυφή των σχετικών πρωτοβουλειών της ελληνικής προεδρίας. Επιδιώκουμε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην ανάδειξη των θετικών πτυχών μιας συνολικής ευρωπαϊκής διαχείρισης του μεταναστευτικού φαινομένου στην υπηρεσία της ανάπτυξης και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναδείξουμε όλες τις διαστάσεις των πολιτικών μετανάστευσης και κινητικότητας με παράλληλες δράσεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την παράνομη μετανάστευση στην οικονομία, την κοινωνική συνοχή και την πολιτική σταθερότητα. Ειδικότερα στον τομέα της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, κύρια προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας θα είναι η νομοθετική προώθηση του νομοθετικού πακέτου για τα έξυπνα σύνορα, για τα smart borders, που όπως γνωρίζετε περιλαμβάνει τρεις προτάσεις κανονισμών. Πρώτον, πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία ενός συστήματος εισόδου-εξόδου, ώστε να καθιερωθεί μητρό στοιχείων εισόδου-εξόδου των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι διασχίζουν τα σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία προγράμματος καταχωρημένων ταξιδιωτών. Και τρίτον, πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού 562 του 2006 όσον αφορά στη χρήση του συστήματος εισόδου-εξόδου και του προγράμματος καταχωρημένων ταξιδιωτών. Επιδίωξη της Ελληνικής Προεδρίας ε, σε σχέση με την πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία συστήματος εισόδου-εξόδου πολιτών τρίτων χωρών είναι η πραγματοποίηση προόδου των συζητήσεων κατά τη δεύτερη ανάγνωση του κειμένου με σκοπό μεταξύ άλλων την εισαγωγή διατάξεων σχετικά με την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου. Όσον αφορά στην πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία προγράμματος καταχωρημένων ταξιδιωτών, θα επιδιώξουμε την ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουν οι συζητήσεις με μια δεύτερη ανάγνωση του κειμένου κανονισμού για τη δημιουργία συστήματος εισόδου-εξόδου πολιτών τριτών χώρων. Ένα άλλο κείμενο που αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την ελληνική Προεδρία ε, αλλά και τόσο για το Συμβούλιο όσο και για το Κοινοβούλιο είναι η πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση κανόνων για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον οργανισμό Frontex. Όπως ξέρετε έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις και έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρεις τεχνικές συναντήσεις. Η Ελληνική Προεδρία θα επιδιώξει την επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση και επιθυμία μας είναι να τα καταφέρουμε πριν από τις ευρωεκλογές. Όπως γνωρίζετε έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση τριλόγου αναφορικά με την πρόταση τροποποίησης των παραρτημάτων του κανονισμού 539 του 2001 που αφορά στην απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης 16 κρατών της Καραϊβικής και του Ειρηνικού των ε, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καθώς και της Κολομβίας και του Περού. Ε, από την πλευρά μας θα ήθελα να διαβεβαιώσω το Κοινοβούλιο ότι η Ελληνική Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί συμφωνία. Σε πρώτη ανάγνωση βέβαια και ε, να υιοθετηθεί ο κανονισμός αυτός πριν πάλι από τις ευρωεκλογέ. Για το σκοπό αυτό και δεδομένων των πιεστικών χρονικών προθεσμιών αποτελεί προτεραιότητα της Προεδρίας μας η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας Συμβουλίου και Κοινοβουλίου έως τις αρχές ε, Φεβρουαρίου και αισιοδοξούμε ότι θα επιτύχουμε στο στόχο αυτό με την στενή συνεργασία όλων. Στο ίδιο πλαίσιο και σε συνέχεια της επιτυχούς εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την απελευθέρωση των θεωρήσεων από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για την μεταφορά της Μολδαβίας στο θετικό κατάλογο του κανονισμού 539 του 2001. Ε, από τη μεριά μας θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την αποδοχή της πρότασης αυτής από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και είμαστε αισιόδοξοι ότι αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες του Κοινοβουλίου θα είμαστε σε θέση να επιτύχουμε μια ταχεία ολοκλήρωση του φακέλου ώστε το συντομότερο δυνατό οι Μολδαβοί πολίτες να δίνανται να ταξιδεύουν στο χώρο Σέγγεν χωρίς θεώρηση. Σε σχέση τώρα με τον τομέα αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικέ υποθέσεις. Στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και σε ό,τι αφορά τις ποινικέ υποθέσεις έχουμε σε εξέλιξη δύο νομοθετικές προτάσεις. Προτάσεις οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους και αναφέρομαι στην πρόταση κανονισμού για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιβολής του Νόμου και τη συγχώνευσή της με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία αλλά και στην πρόταση κανονισμού για τη μεταφορά της έδρας της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. Για την Ελληνική Προεδρία η αναβάθμιση της Europol ε, είναι ένας πολύ σημαντικός φάκελος ε, που υπόκειται σε ό,τι προβλέπεται από τη διαδικασία της συνθήκης της Λισαβόνας και επηρεάζει φυσικά τον πυρήνα της συνεργασίας των αρχών εφαρμογής του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης εν γέννη. Θα ήθελα να ε, ε, σας ενημερώσω ότι η εξέταση της πρότασης κανονισμού σε επίπεδο ομάδας εργασίας είναι εν εξελίξη από τον Ιούνιο του 2013 και από την πλευρά μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προωθήσουμε το φάκελο μέχρι το τέλος της Προεδρίας μας υιοθετώντα τη θέση του Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση του Ιουνίου. Πέραν του κανονισμού για τη Europol, θα ήθελα να αναφερθώ και στην πρόταση κανονισμού για την έδρα της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, της ΕΠΟΛ. Όπως γνωρίζετε, δεδομένης της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να μην φιλοξενήσει πλέον την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, το Συμβούλιο αποφάσισε τον Οκτώβριο να μεταφερθεί η έδρα της Ακαδημίας στην Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία. Προς τούτο, τον περασμένο Νοέμβριο, 25 κράτη-μέλη παρουσίασαν μια νομοθετική πρωτοβουλία για την τροποποίηση της απόφασης για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Ε, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι έχετε ήδη ορίσει συγκητή για το συγκεκριμένο θέμα και να σας ενημερώσω ότι στηριζόμαστε απόλυτα στη συνεργασία σας ώστε λόγω του κατεπήγοντος του θέματος να επιτύχουμε την υιοθέτηση νομοθετικής πρωτοβουλίας πριν από τις ευρωεκλογέ. Πιστεύω ότι αποτελεί κοινό μας ε, συμφέρον και κοινό μας στόχο να διατηρήσουμε επιχειρησιακή την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Σε σχέση τώρα με, την, με το μέλλον, με τη μελλοντική ανάπτυξη του τομέα δικαιοσύνης εσωτερικών και εσωτερικών υποθέσεων. Όπως γνωρίζετε, σε εκτέλεση των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2013, το Συμβούλιο θα καταρτήσει τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για το νομοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό για τον τομέα ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας που θα έρθει ε, να αντικαταστήσει, να διαδεχθεί ακόμα καλύτερα το υφιστάμενο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Ως ελληνική προεδρία θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε όλους ότι θα συνεργαστούμε στενά με τα κράτη-μέλη αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την οποία περιμένουμε την έγκαιρη συμβολή της με την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης το Μάρτιο. Παράλληλα θα επιδιώξουμε την ενεργή συμβολή του έτερου ε, συνομοθέτη, ε, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο θα κληθεί να υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2014, να ανταποκρίνεται στις πραγματικές μελλοντικέ ανάγκες του τομέα ΔΕΗ. Στο ανωτέρο πλαίσιο, το μέλλον του τομέα ΔΕΗ θα απασχολήσει την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων, η οποία θα προετοιμάσει και τις περαιτέρω ε, συζητήσεις. Okay. Θα τελειώνω. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διαξοδικό στο θέμα κατά το άτυπο Συμβούλιο ΔΕΗ ε, στην Αθήνα 23 και 24 Ιανουαρίου ε, με τη συμμετοχή και των εκπροσώπων των Επιτροπών ΛΥΜΠΕ και Γιούρι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με αυτά Ελπίζω να μην σας κούρασα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε τον λόγο. Thank you. No. Ευχαριστώ. Ας προχωρήσουμε. Let's, let's make our best to fill in the timing up until 5.30, which is... Έχουμε χρόνο μέχρι τις 5.30. Ας αξιοποιήσουμε αυτό το χρόνο να μιλήσουν οι επόμενοι ευρωβουλευτές. Ο κύριος Παπα-Νικολάου είναι πρώτος. Thank you, thank you very much, Mr. Mr. President. I will... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω ελληνικά, για να τιμήσω και την Προεδρία μας. Ε, θα αισθάνομαι και πιο άνετα εξάλλου μπροστά στου Έλληνε υπουργού. Κύριε Υπουργέ των Ιστορικών, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Γεωργιάδη, για την εισαγωγική σα τοποθέτηση για την ελληνική προεδρία. Είχαμε συνεννοηθεί προηγουμένω με την κυρία Ματιέ να κάνω εγώ έτσι την πρώτη εισαγωγή για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για να σα καλωσορίσουμε. Το έκανε η κυρία Ματιέ. Ε, ήθελα να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση μετά από όσα ακούστηκαν όμω και την πρώτη απάντηση των ε, την πρώτη δική σας απάντηση και τις ερωτήσεις των συναδέλφων θέλω να, να, να, κάνω μια πιο εξειδικευμένη τοποθέτηση. Άκουσα με πολύ προσοχή αυτό που είπε η κυρία Βερζιά, δεν ξέρω αν είναι ακόμη εδώ η κυρία Βερζιά είναι μια από τις, ξέρετε μετά από τόσα χρόνια, ειδικά σε μια επιτροπή όπως η ΛΥΜΠΕ, που είχαμε έτσι πολύ έντονες στιγμές και είναι μια επιτροπή που οι αντιθέσεις είναι πολλές φορές μεγάλες και με πολύ κόπο φτάνουμε σε συνθέσεις και αποφάσεις. Ε, η κυρία Βερζιά είναι μια από εκείνες συναδέλφου που ανήκει στην ομάδα της ΓΚΟΕ αλλά πάντα με πολύ καθαρή τοποθέτηση, ε, αντιλαμβάνεται τα μηνύματα και είναι πάντα αντικειμενική στην παραστήρισή της και στην αξιολόγηση των πραγμάτων. Ε, ήθελα λοιπόν να της πω, αλλά δεν είναι εδώ δυστυχώς ελπίζω να της μεταφερθεί αυτό που θα της πω, ότι ναι μεν υπάρχουν πάντα οι NGOs οι οποίοι μεταφέρουν κάποια μηνύματα για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, την ίδια στιγμή όμως θα ήθελα και εγώ να ζητήσω λίγο χρόνο από εκείνη για να της, ή εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, για να τη μεταφέρω την προσπάθεια που το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές εδώ στην Επιτροπή μας και το καλοκαίρι ήταν εδώ και ο κύριο Ζένδιας, ο αρμόδιος υπουργό, σε σχέση με τη νέα υπηρεσία ασύλου που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα, σε σχέση με τα νέα κέντρα υποδοχής που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα, σε σχέση με την αυξημένη προστασία πλέον που έχουν όλοι όσοι εισέρχονται στη χώρα, σε σχέση με την αυξημένη φύλαξη των συνόρων και τις εκθέσεις του Σέγγεν που έχουμε πλέον, οι οποίες επιχαίρουν για την προσπάθεια της Ελλάδας, σε σχέση με τα σχόλια της ΕΑΖΟ ότι η Ελλάδα πλέον διαθέτει τους πιο καταρτισμένους υπαλλήλους στον τομέα των υπηρεσιών ασύλου. Αυτά θα ήθελα έτσι να τα κουβεντιάσω και εγώ πριν κανείς βγάλει συμπεράσματα και στα πλαίσια μιας προεδρίας που προέρχεται από την Ελλάδα μετά από τόσο, δύσκολες, από τόσο δύσκολη περίοδο που έχει περάσει και μέσα στην κρίση έχουμε μια Προεδρία πραγματικά προσπαθεί που νομίζω βλέπουμε ότι είναι πραγματικά προετοιμασμένη σε όλα. Είναι κρίμα να υιοθετούμε μονομερώς κάποιες απόψεις. Ξέρετε πάρα πολλά ότι ε, και όλοι μας εδώ και όλοι οι συνάδελφοι από το EPP Group πάντα δίνουμε την μεγαλύτερη έμφαση είναι απόλυτη προτεραιότητα ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων. Κανείς δεν δέχεται καμία έκπτωση. Όμως να βλέπουμε, ε, αν μπορώ να το παρακαλέσω αυτό, ισορροπημένα τα πράγματα. Ε, κύριε Υπουργή, η, ερώτησή μου είναι απλή και δεν θέλω να, να κάνω κατάχρηση του χρόνου. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε κουβεντιάσει στα θέματα της πολιτικής ασύλου και της μετανάστευσης. Αυτό θα εστιάσω γιατί πριν ερωτήθηκαν ο κύριος Μιχελάκης, ο κύριος Αθανάσιο και οι άλλα θέματα. Έχουμε, έχουμε εστιάσει, αλλά θα ήθελα και από τον κύριο Μιχελάκη μια απάντηση, γιατί στον τομέα της νόμιμη μετανάστευσης είναι εκείνος αρμόδιος. Έχουμε κουβεντιάσει για το θέμα της δίκαιης κατανομής των βαρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη αλληλεγγύη που σε πραγματικό επίπεδο πρέπει να, να, να υιοθετήσουμε, να την αυξημένη ε, ε, αλληλεγγύη που χρειαζόμαστε ιδιαίτερα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που δέχονται το μεγαλύτερο μέγεθος των, των ροών των μεταναστών από τις γειτονικές μας χώρες που πραγματικά εκεί υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Αισθάνεστε ότι τα καταφέραμε αυτή την περίοδο. Η ελληνική προεδρία που είναι μια προεδρία που έρχεται να κλείσει και τη δική μας θητεία που έρχεται πριν από τις εκλογές. Με την έμφαση που θέλει να δώσει τη μετανάστευση σκοπεύει να πει περισσότερα για τα θέματα αυτά. Το πρόγραμμα εσωτερικής μετεγκατάστασης μεταναστών, το Relocation Program, θα μπορέσει να προωθηθεί κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας και νομίζω αυτό συμφωνούμε όλες οι πολιτικές ομάδες. Το ζήτημα της κατανομής των βαρών, όχι μόνο στην, στις ροές των μεταναστών αλλά και, στην, και στον τομέα του ασύλου και στον τομέα των ευθυνών πρέπει να έχουμε σκεπτόμαστε να το δούμε ακόμη πιο προωθημένα και να πείσουμε έτσι τους Ευρωπαίους πολίτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της αναλαμβάνει την ευθύνη γιατί ξέρετε σήμερα υπάρχει μια αίσθηση ότι άλλες χώρες πιέζονται περισσότερο, άλλες λιγότερο. Υπάρχουν επιμέρους επιχειρήματα και διαφορετικές προσεγγίσεις. Εν πάση περιπτώσει όλοι νομίζω συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη αλληλεγγύη. Και θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο για το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Sorry for the abuse of time, Mr. President. Συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου, κύριε Πρόεδρε. Thank you, Mr. Σας ευχαριστούμε κύριε Παπα-Νικολάου. Κύριε Κάσμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Κύριε Μιχελάκη, να σας ευχαριστήσω για την ε, παρουσίασή σας και το πάθος σας. Προέρχομαι από το Ηνωμένο Βασίλειο και πιστεύω πως όλες οι χώρες έχουν πληγεί από τον εξτρεμισμό που προκάλεσε η οικονομική κρίση. Δεν νομίζω λοιπόν πως χρειάζεται εμεί να κάνουμε διάλεξη στην Ελλάδα για δικαιώματα για ε, την άνοδο του εξτρεμισμού και για παραβιάσεις δικαιωμάτων. Είναι κάτι που ζούμε και στις χώρες μας. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά και το βλέπουμε και στην περίπτωση της χρήση αυγή. Να ε, δώσουμε όμως και τα εύσημα στην, ε, στους Έλληνες, γιατί επέζησαν από αυτήν την κρίση. Και η κρίση προέκυψε λόγω έλλειψης ηγεσία σε υπουργικό επίπεδο, σε επίπεδο αρχηγών ε, κρατών, κυβερνήσεων στα κράτη-μέλη. Και πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ως ε, εισηγητής λοιπόν ε, τη αναθεώρηση του κανονισμού 1049, θα ήθελα να σας μεταφέρω την άποψη ότι τα θέματα δεν είναι τεχνικής φύσεως, ούτε και τα προβλήματα είναι τεχνικά. Στο επίπεδο του Συμβουλίου υπάρχει έλλειψη πολιτικής θέλησης και άρχισε από την Δανική Προεδρία το συνέχισε η Λιθουανική Προεδρία, όμως ε, αυτό το ζήτημα μπλοκάρεται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν ε, να σας δείσω να δώσετε τη δέουσα προσοχή, διότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς τους πολίτες και ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών. Αυτή η άνοδος των ε, ακραίων κομμάτων είναι επικίνδυνη. Χρειάζεται επίσης να προωθηθεί στο Συμβούλιο η καταπολέμηση των διακρίσεων και ο κανονισμός κατά των διακρίσεων. Είναι τα θεμέλια οποιασδήποτε πολιτισμένης κοινωνίας και ιδιαίτερα κράτους μέλους και οποιοδήποτε άμεσα εκλεγμένου κοινοβουλίου. Και τέλος, να σας πω ότι οι ανησυχίες που εκφράστηκαν για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ομοφιλοφίλων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κρίσης είναι κάτι που μας ε, ανέφεραν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που είναι βασισμένες στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διεθνώς. Και γι' αυτό το αναφέρω, όμως ε, ξανά κύριε Μιχελάκη θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι μιλήσατε για την ουσία των πραγμάτων χωρίς κομματικές αποχρώσεις. Εάν πραγματικά θέλουμε οικονομική ανάπτυξη, πρέπει να δώσουμε κοινωνική δικαιοσύνη. Το ένα πάει μαζί με το άλλο. Κύριε Κάσμαν, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Λάντφορντ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς ε, όλους εσάς. Ήθελα και εγώ να αναφέρω το θέμα των ανθρωπινών δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Αύριο έχουμε μία παρουσίαση για τα εγκλήματα μίσους από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τον ΦΡΑ, και σίγουρα δεν υποτιμώ την πρόκληση που αντιμετωπίζει η χώρα σας και η Προεδρία σας. Αλλά βασίζομαι και εγώ στις πληροφορίες που λαμβάνω από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και χωρίς να παραγνωρίζω την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τις προσπάθειες που γίνονται από την παρούσα κυβέρνηση για την καταπολέμηση της βίας, η αλήθεια είναι ότι έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις χωρίς σχεδόν καμία δίωξη και καμία καταδίκη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο που σχετίζεται με την απόφαση πλαίσιο του 2008 και την ενσωμάτωσή της για, την, για τα εγκλήματα μίσους και τα ρατσιστικά εγκλήματα. Μπορείτε εσείς να μας διαβεβαιώσετε ότι θα υπάρξουν προσπάθειες στο νομοσχέδιο αυτό να ενισχυθούν τα σημεία αυτά στην ελληνική νομοθεσία που αντιμετωπίζουν και καταπολεμούν τα εγκλήματα μίσους, ρατσισμού και να αξιοποιήσουν τις μέγιστες δυνατές ποινές για αυτά τα εγκλήματα. Το πρόστιμο, αν δεν κάνω λάθος, είναι πόσο, 100 ευρώ. Και αν δεν κάνω λάθος, 100 ευρώ πρέπει να δώσει κάποιος για να καταθέσει μήνυση. Μπορείτε να μας πείτε επίσης τι, τι θα γίνει με την περίπτωση των παράνομων μεταναστών που είναι θύματα τέτοιων εγκλημάτων. Και επίσης υπάρχει κάποια κατάρτιση που προβλέπεται για τους αστυνομικούς ώστε να, και τους εισαγγελείς ώστε να αντιμετωπίζουν αυτά τα φαινόμενα. Επίσης, μια που ανέφερα την αστυνομία, ε, θα ήθελα να αναφερθώ στην επιχείρηση Ξένιος Δίας. Και ο κύριος Παπα-Νικολάου ανέφερε κιόλας ότι υπάρχει συμπεριφορά ε, ρατσιστική και με διακρίσεις της αστυνομίας, ότι σταματούν μετανάστες στο δρόμο χωρίς βάσιμες υποψίες, χωρίς κανένα λόγο. και το 6% των ε, ανθρώπων που σταματούν στο δρόμο οι αστυνομικοί ε, είναι άνθρωποι που δεν, ε, δεν έχουν δώσει καμία, κανένα δικαίωμα για υποψίες. Υπάρχει λοιπόν κάποια πρόβλεψη, υπάρχουν κάποιες ε, κατευθυντήριες γραμμές του τι γίνεται. Υπάρχει κάποια πρόθεση να αλλάξουν αυτές οι πρακτικές και αυτή η συμπεριφορά. Αυτό το ρωτάω διότι έχετε την Προεδρία και, θέλω, και ξέρω πως θέλετε να ε, επιτευχθεί πρόοδος για αυτά τα θέματα, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Έρνστ. Σας ευχαριστώ. Θα μεταφέρω και εγώ στους συναδέλφους μου τους ευγενικούς χαιρετισμούς του κυρίου Παπα-Νικολάου. Να σας ε, ρωτήσω το εξή. Αναφέρετε ω προτεραιότητά σα στην πολιτική ασύλου, ασύλου και μετανάστευσης. Μας ε, αναφέρετε και μερικά νούμερα, τα οποία πραγματικά, έτσι όπως τα παρουσιάσατε, είναι κάτι που πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ στα σοβαρά. Υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγες, ε, μετανάστες, ε, είτε νόμιμοι είτε παράνομοι στην Ελλάδα. Όντω. όμως έχουμε ένα πακέτο για το άσυλο εδώ. Και στο πακέτο αυτό δεν αναφέρεται ούτε οι, ούτε οι αρμοδιότητες, ούτε προβλέπετε κάτι για τους ετούντες άσυλο. Εσείς τι προτίθεστε να κάνετε για το πακέτο του ασύλου. Το πρόβλημα, το κύριο πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό στην ουσία. Και αυτό θεωρώ πως είναι πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά το άσυλο επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν προβλέπονται βελτιώσεις, αν υπάρχει ε, κάποια βελτίωση. Πραγματικά είναι άσχημη η κατάσταση στην Ελλάδα. Ξέρετε τι κριτική έχει ασκηθεί στην ε, διαδικασία. Ξέρετε τι αποφάσεις έχουν ληφθεί από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μπορείτε εσείς να ε, διασφαλίσετε, να εγγυηθείτε ότι θα υπάρχουν καλές συνθήκες στις ε, συλλήψεις, στις κρατήσεις των ε, μεταναστών αυτών. Έπειτα, οι κατευθυντήρες γραμμές για τα θαλάσσια σύνορα. Αναφέρθηκε το θέμα αυτό ήδη από κάποιον συνάδελφο. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη τοποθετηθεί για αυτό το θέμα. Έχουμε και τη σχετική έκθεση που έχει ήδη υποβληθεί. Τι γίνεται όμως στο Συμβούλιο με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα θαλάσσια σύνορα. Τι ενέργειες σκοπεύετε να κάνετε. Έπειτα, έξυπνα σύνορα. Είχαμε ήδη κάνει μια ακρόαση που νομίζω ο κύριος Κοέλιο είχε ρωτήσει για το κόστος. Πόσο κοστίζει αυτό το σύστημα καταχώρησης εισόδου-εξόδου. Υπάρχουν κάποιες προβλέψεις γι' αυτό. Και αυτό θα ήταν κάτι που θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Τέλος, αναφέρεται το δεξιό εξτρεμισμό ε, με συνέστημα. Και μας είπατε ότι υπάρχει σύνδεση αυτού του φαινομένου με την οικονομική κατάσταση, με την ένδια. Φυσικά και η Ελλάδα δεν είναι ακροδεξιά χώρα. Όμως δεν νομίζετε πως η πολιτική λιτότητας η οποία έχει οδηγήσει σε αυτή την καταστροφή είναι κάτι που έχει συμβάλει στη δημιουργία αυτής της άσχημης κατάστασης της ακροδεξιάς. Και, αυτό, και αυτή η πολιτική ήταν κάτι που έχει στηρίξει η κυβέρνησή σα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπρόνς. Θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση που θα κάνω τώρα στον Υπουργό Δικαιοσύνη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αλλά φυσικά προηγούνται οι συντονιστέ στη ΛΥΜΠΕ. Είμαστε όλοι ίσοι, αλλά κάποιοι είναι πιο ίσοι από του άλλου. <clears throat> θα το ρωτούσα λοιπόν, εάν κατά τη διάρκεια τη ελληνική προεδρία έμαθε ότι ένα άλλο κρατος μέλος είχε ε, συλλάβει διάφορους βουλευτές μετά από μια πολιτική δολοφονία ενός ακτιβιστή. Αυτός που συνελήφθη όμως, αν ας πούμε δεν είχε κατηγορηθεί, αν δεν υπήρχαν στοιχεία για την ανάμειξή του, ποια θα ήταν η αντίδρασή σας. Και αν, α πούμε, μετά από αυτή τη δολοφονία το αποτέλεσμα ήταν δύο άλλε ιδεχθεί δολοφονίε. Αν οι βουλευτές διαπράττουν κάποιο αδίκημα, βεβαίως πρέπει να διώκονται. Θα πρέπει να είναι και αυτοί εξίσου ένοχοι, όχι λιγότερο ένοχοι. Συμφωνείτε ότι η σύλληψη πολιτικών και βουλευτών ειδικά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με σκεπτικισμό ως προς την προσέγγιση που πρέπει να έχουμε. Η θέση όμως το... και η πολιτική τοποθέτηση αυτών των βουλευτών θα πρέπει να είναι άσχετη με το αν θα διωχθούν ή όχι. Όμως αυτό δεν φαίνεται από τη σημερινή συζήτηση. Γιατί έχει έτσι μια απόχρωση η σημερινή συζήτηση που μας θυμίζει α, ότι μιλάμε και κολλάμε συνέχεια σε θέματα όπως ακροδεξιά κτλ. Ε, έχει έτσι μια χρειά ιδιαίτερη η σημερινή συζήτηση. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Ο κύριος Μέλλο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τον Υπουργό Εσωτερικών. Θα ήθελα να πω σύντομα το εξή. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση της ζωής της Ευρώπης, αυτό που θα πρέπει να μας ανησυχεί είναι η ανάδυση κάποιων ε, ε, εξτρεμιστών, εξτρεμισμών κάθε είδους, εξτρεμισμών άκρας δεξιάς ή άκρας αριστεράς. Είδαμε να ξαναζούν ε, φαινόμενα όπως αυτοί που πολιτικά είναι κατά του ΝΑΤΟ, κατά του ευρώ, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όλος παραδόξως εκλέγονται για να ασκήσουν μάλιστα και καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία δεν συμπαθούμε. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, μέσα από την προπτική κάποιου που παρακολουθεί από την Νότια Ευρώπη, την Ιβυρική Χερσόνησο. Η Ελλάδα λοιπόν έχει ζήσει και τα δύο είδη εξτρεμισμού πρόσφατα, και την άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά. Και όλο ένα αυξάνονται οι ανησυχίες και προσθέτω ότι το παρακολουθώ όλα αυτά με πολύ ανησυχία γιατί είδαμε εδρεωμένα δημοκρατικά κόμματα που για χρόνια εναλλάσσονταν στην εξουσία στην Ελλάδα, απελευθέρωσαν ένα κομμάτι του πολιτικού χώρου λόγω των συγκυριών που επικρατούν στη χώρα και καταλήφθηκαν από κόμματα της άκρης δεξιάς και της άκρης αριστεράς. Και νομίζω πως με όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, εγώ πιστεύω σε μια Ευρώπη που αποτελείται από αλληλεγγύη και συνοχή. Η άκρα δεξιά και η άκρα αριστερά σημαίνουν διχασμό, διχόνοια και εγωισμό. Και επειδή η Ελλάδα ζει αυτό το φαινόμενο, καθημερινά με ποιο τρόπο η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσει να καταβάλει μια τέτοια προσπάθεια που να έχει και κάπως παιδαγωγικό χαρακτήρα έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει άλλους δρόμους, να μπορέσει να καταπολεμήσει όλες αυτές τις ακρότητες και να έχετε υπόψη σας κύριε Υπουργέ ότι όλα αυτά όλα αυτά θα πρέπει, μπορούν να γίνουν καλύτερα μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο έχουμε ευρωβουλευτές που αντιπροσωπεύουν κόμματα τα οποία, ε, αν και είναι λίγοι, στις δικές τους χώρες ε, υποστήριξαν ε, να γίνουν γενετικά τεστ ώστε να εξακριβωθεί εάν οι εκπρόσωποι τους είχαν εβραϊκό αίμα. Ένα σκάνδαλο λοιπόν αντισημιτικό το οποίο μας ντροπιάζει όλους. Αυτή είναι μια φάση εξτρεμισμού που θυμίζει το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και αυτό έγινε τώρα, σήμερα, δηλαδή αυτή την εποχή. Η Ελλάδα λοιπόν στην Προεδρία μπορεί να ασκήσει έναν παιδαγωγικό ρόλο ώστε η Ευρώπη να ξαναγυρίσει στο σωστό δρόμο και να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Ρομέρο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σε σχέση με την Τουρκία και την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Αυτή την εβδομάδα θα μιλήσουμε στο Κοινοβούλιο για συμφωνίες επανεισδοχής και για τις ιδιαίτερες σχέσεις και συμφωνίες με την Τουρκία. η οποία δεν απαιτεί θεώρηση για διαβατηρίων για τους επισκέπτες. Εσείς, ε, εγώ πιστεύω ότι είναι πρόβλημα αυτό. Εσείς τι πιστεύετε και έπειτα, Γιατί κατά τη γνώμη σας το καθεστώς πρόσφυγα δίνεται τόσο λίγο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες του Νότου, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα. Αυτό συνδέεται με το κανονισμό του Δουβλίνου. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το κανονισμό που θεωρητικός δημιουργήθηκε για να αποφευθούν οι απάτες, αλλά δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι για να απεφευθούν οι απάτες πέρα από τον κανονισμό του Δουβλίνου. Ε, και το τελευταίο μου ερώτημα δεν έχει καμία σχέση με τη μετανάστευση, αλλά περισσότερο έχει σχέση με το πακέτο για την προστασία των δεδομένων. Πιστεύετε πως αυτό το πακέτο θα εγκριθεί μέχρι το τέλος της θητείας και μπορείτε να ζητήσετε από το Συμβούλιο να αντιδράσει άμεσα για το θέμα αυτό. Πρόεδρος, ο κύριος Χρυσόγελος. Σας ευχαριστώ. Ε, <clears throat> πολλές φορές ο ρατσισμός πατάει σε μια προϋπάρχουσα στην κοινωνία αντίληψη ότι οι μετανάστες φέρνουν όλα τα κακά, όπως και η ελεύθερη μετακίνηση, μετακίνηση εργαζομένων. Πάνω σε αυτοί έρχονται να κερδοσκοπήσουν εκλογικά ακροδεξιά κόμματα. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί οι χώρες όπως είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, υποφελήθηκαν από τη μετανάστευση. Περιμένουμε λοιπόν εμεί από την ελληνική προεδρία που έχει ζήσει και το φαινόμενο τη μετανάστευση να αναδείξει τα θετικά στοιχεία τη μετανάστευση, μετανάστευσης, ιδιαίτερα πρώτων εκλογών. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλε οι έρευνε στην Ελλάδα δείχνουν ότι οι μετανάστες συνεισφέρουν 1% στο ΑΕΠ. Δεν αφαιρούν από το ΑΕΠ, προσφέρουν στο ΑΕΠ. Το ίδιο ισχύει σε πολλέ άλλε χώρε. Περιμένουμε λοιπόν στα πλαίσια τη θεματική προτεραιότητα για τη μετανάστευση που έχετε βάλει ότι είναι ένα από τα πέντε θέματα ω Προεδρία σε όλη την Ευρώπη να γίνει μια μεγάλη καμπάνια για το πώ έχουν επιφεληθεί οι χώρε και οικονομικά. Εάν λέμε συνέχεια ότι η μετανάστευση είναι βάρο, προφανώ μετά έρχονται οι ακροδεξιοί και λένε αφού είναι βάρο να του διώξουμε. Όλα όμω τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι συνεισφέρουν οικονομικά και κοινωνικά και στα ασφαλιστικά συστήματα και πολλέ χώρε ε, εποφελούνται, ζητάνε να έρχονται μετανάστες. Άρα περιμένουμε από την Προεδρία να αναδείξει αυτό το θέμα. Το δεύτερο είναι το πρόβλημα, μιλάμε πολύ συχνά για μετανάστες που είναι παράνομοι, που δεν έχουν χαρτιά. Υπάρχουν νόμιμοι δρόμοι μετανάστευση σήμερα μέσω της Ελλάδας. Δεν υπάρχουν νόμιμοι δρόμοι. Άρα προφανώς όποιος έρχεται, ακόμα και Σύριος πρόσφυγας, είναι παράνομος. Ξέρετε ότι πολλά από τα θύματα σήμερα είναι Σύριοι πρόσφυγες. Εννιά άτομα βρήκαν το θάνατο χτες, αν δεν κάνω λάθος, στο Αγαθονήσι και είναι παιδιά. Έχουν βρει το θάνατο πολλοί από τους 177 ετησίως που πεθαίνουν 180-200 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πολλοί από αυτούς προσπαθούν να επανενωθούν με οικογένειες στην Ευρώπη. Υπάρχουν, είναι γονείς που ζουν στην Ευρώπη, φέρνουν τα παιδιά τους, ε, οι γυναίκες να βρουν τους άντρες τους. Εάν μειώσουμε λοιπόν όλο αυτό το ποσοστό, θα δείτε ότι το 20-30% είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί βασανιστήρια. Είναι άνθρωποι που θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Άρα τα νούμερα δεν δείχνουν την εικόνα, είναι πολύ λιγότεροι γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν την προστασία των ανθρώπων που δικαιούνται άσυλο ή που δικαιούνται να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Λοιπόν, περιμένουμε η Ελλάδα και οι άλλες περιοχές να έχουν κέντρα υποδοχής ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα τι γίνεται. Και το τρίτο είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Πάρα πολλά λεφτά πάνε στην προστασία των συνόρων. Απλώς μετακινούν τα παράνομα κυκλώματα σε κάποια άλλα σημεία. Είπατε και σωστά ότι μειώνεται η είσοδος από τον Εύρο, αλλά μεταφέρεται η είσοδος από άλλες περιοχές, από νησιά, πιο κάτω, στο Νότιο Αιγαίο, στη Λαμπετούσα κλπ. Δεν μπορούμε να έχουμε πολιτική που δίνει τα περισσότερα χρήματα και όλη την προσπάθεια στο να αποτρέψει. Πρέπει να έχουμε πολιτική νόμιμης εισόδου και πολιτική που ενισχύει την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Προφανώς αν είναι οι άνθρωποι χωρίς δικαιώματα πεταμένοι σε μια πλατεία θα δημιουργούν προβλήματα, ενώ αν υπάρχουν πολιτικές ένταξεις είναι αλλιώς η αντιμετώπιση. Τότε ενσωματώνονται στην οικονομία, στην κοινωνική ζωή, μπορεί να αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης. Και είναι πολύ κρίσιμο πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα όλοι στην Ευρώπη ενώπιση των ευρωπαϊκών εκλογών. Όλη η ακροδεξιά στοχεύει και χρησιμοποιεί αυτό το φόβο απέναντι στον διαφορετικό. Α δείξουμε ότι ένα άνθρωπο σαν και εμά ότι αν έχουμε καλύτερη πολιτική ευρωπαϊκή θα ενσωματωθούν καλύτερα στι κοινωνίε ευρωπαϊκέ και δεν υπάρχει κανένα λόγο να καλλιεργούμε το ρατσισμό γιατί στρέφεται και ενάντια στους πολίτε ευρωπαϊκή καταγωγή που και αυτοί πηγαίνουν σε άλλε χώρε. Έτσι δεν είναι. Στην Αυστραλία, στην Αμερική και μέσα στην Ευρώπη μετακινούνται οι άνθρωποι. Το ίδιο παιχνίδι παίζεται και με, τους, με την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων. Βγαίνει ο, προ, Πρωθυπουργό της Βρετανίας και λέει ότι η ελεύθερη μετακίνηση θα καταστρέψει το κοινωνικό σύστημα της Βρετανίας. Έχουμε και πρόβλημα χρόνου. Έχουμε πίεση χρόνου. Έχουμε τον κύριο Τούσα ο οποίο θέλει και αυτό να κάνει κάποιε ερωτήσει. Παρακαλώ όμω αυτό περιοριστείτε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και έχουμε άλλα δύο σημεία πριν να ολοκληρώσουμε τη σημερινή συνεδρίαση στι 6.30. Κύριε Τούσα. Αντιλαμβάνομαι εκεί που επικεντρώθηκε η συζήτηση, στο σκέλος ε, που παρακολούθησα, είναι στο άσυλο και στη μετανάστευση. Είναι ένα σοβαρό, μεγάλο πολιτικό ζήτημα που δεν έχει να κάνει μόνο με τις χώρες που βρίσκονται περιφερειακά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι συνολικά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου να κάνω μια εκτίμηση που είναι του κόμματός μου βασική. Ό,τι μέτρα και αν παρθούν επιμέρους σε ό,τι αφορά τον περιορισμό εισόδου προσφύγων και μεταναστών από τρίτες χώρες δεν θα έχουν αποτέλεσμα και αν ακόμα θέλετε στρατιωτικοποιηθεί ακόμα περισσότερο η Frontex, αν ακόμα ενισχυθεί και δημιουργηθεί ευρωπαϊκή ακτοφυλακή, αν σηκωθούν ακόμα τύχη μεταξύ των κρατών μελών, όταν ο άλλος στο σπίτι του, στη γειτονιά του νιώθει τις βόμβες να διαλύουν την οικογένειά του, τους δικούς τους ανθρώπους θα ανατρέξει σε μία λύση. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτοί που βρίσκουν 4 και 5 χιλιάδες ευρώ για να δώσουν στους δουλέμπορους για να μετακινηθούν μέσα από αυτό τον παράνομο μηχανισμό που απομισά δισεκατομμύρια δολάρια δεν είναι οι πιο πλούσιοι. Είναι αυτά τα στρώματα, τα μεσία τα στρώματα που κάπως είχαν οργανώσει με ένα ανεκτό τρόπο στη χώρα τους να ζήσουν τη ζωή τους. Κανένας δεν φεύγει από τη χώρα του γιατί έτσι θέλω. Για πέστε μου σας παρακαλώ. Μπορεί πραγματικά να ανακοπεί αυτό το κύμα των ροών των μετανοστών όταν χθε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίστηκε να σταθεί εξατευτικό σώμα στην κεντροαφρικανική δημοκρατία εχωρώντας το στρατηγείο της Λάρισας για το σχεδιασμό και την οργάνωση αυτής της στρατιωτικής αποστολής. Δηλαδή, θεωρούμε ότι τέτοιες αποφάσεις μπορούν να ανακόψουν αυτά τα στρατιωτικά ρεύματα. Θα επιβάλλουν την ειρήνη μεταξύ των αντιμαχόμενων ομάδων. Αυτό έγινε στο Μάλι. Αυτό έγινε στη Λιβύη. Αυτό έγινε στη Συρία μακριά από μας η δεοληψία ε, είναι ένα ζήτημα. Θα παραμείνει ο κανονισμός του Βιβλίνο 2 και στη συνέχεια έτσι να παραμένουν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες εγκλωβισμένοι χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγοι και πρόσφυγες. Θα παραμένει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση και με αυτό τελειώνω. 16, κάτω από 16 χρονών παιδιά μεταναστών επειδή μπήκαν με τους γονείς τους. Ιστάθηκαν από τους γονείς τους και συνελήθηκαν. Να πηγαίνουν στη φυλακή μέχρι και 18 μήνες. Θα συνεχίσουμε να λέμε, ξέρετε κάτι, ε, τα, κέντρα, ε, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες με απαράδεκτες συνθήκες ε, ζωής λέγονται κέντρα φιλοξενίας. Δεν θέλω να λαϊκής και το είναι επιτρεπτό ούτε από το κόμμα μας έχουμε αυτή την ε, επιλογή. Είναι σοβαρό, σοβαρότατο πολιτικό ζήτημα. Και να κλείσω με το εξή, επιτρέψτε μου. Όσοι προσπάθησαν, ναι κύριε Πρόεδρε, κατανοώ και ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Όσοι προσπάθησαν να ποινικοποιήσουν την ιδεολογική και πολιτική δράση των κομμάτων φούσκωσαν τα πανιά των φασιστικών ναζιστικών οργανώσεων παρόμοιων της χρυσή Αυγής κριτής ολονών μας είναι ο λαός στις χώρες που εκλεγόμαστε. Ας μην υποτιμούμε ούτε τη μνήμη ούτε την κρίση τους. Ευχαριστώ. Thank you. you we're running out of time. It's been a huge round of questions. Είχαμε ακούσει πολλές ερωτήσεις, δεν έχουμε πολύ χρόνο και πρέπει να απαντήσουν και οι υπουργοί. Κύριε Ποτασίεβιτς, ζητάτε το λόγο, αλλά προσπαθήστε να μην ε, μιλήσετε για πέντε λεφτά, γιατί αλλιώς έχουμε πρόβλημα, δεν θα προλάβουμε να διεκπαιρεώσουμε και τα υπόλοιπα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Πρέπει και αυτά να τα κοιτάξουμε πριν τις 6.30. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο Ε, θα μιλήσω πολωνικά όμως. Δεν θα μιλήσω για πέντε λεφτά, πολύ λιγότερο. Ως εισηγητής για την οδηγία είμαι ικανοποιημένος που η Ελληνική Προεδρία ανταποκρίθηκε και τη θεωρεί αυτή την οδηγία προτεραιότητά της. Το θέμα των ναρκωτικών είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και χαίρομαι που αντιμετωπίζετε με πολύ σοβαρότητα την οδηγία αυτή και την έχετε βάλει στις προτεραιότητές σας. Εγώ επίσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δουλεύω για θέματα ανατολική γειτονία και χαίρομαι που η Ελληνική Προεδρία θέλει να απελευθερώσει από την υποχρέωση ε, θεωρήσεων τους πολίτες της Μολδαβίας μέχρι το τέλος της θητεία τη. Για το σύστημα διαχείρισης των μεταναστών πιστεύω ότι θα βρούμε μια λογική λύση. Έχουμε, Έχουμε λοιπόν λίγα λεπτά. Πρότεινα λοιπόν να απαντήσει στην αρχή πρώτος ο κύριος Μιχελάκης και μετά ο κύριος Γεωργιάδης. Κύριε Μιχελάκη, θα ήθελατε να αρχίσετε. Εκτός μικροφώνου. Μάλιστα. Αν θέλετε λοιπόν να αρχίσετε πρώτος, παρακαλώ. Και μετά θα ακούσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριε Γεωργιάδη. Precisely, that's what I said, Mr. Αυτό ακριβώς είπα. Κύριε Μιχελάκη, αρχίστε. Καθαρίσαμε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν ε, πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν. Πιστεύω ότι έχει γίνει ένας γόνιμος διάλογος και έχουν ακουστεί πάρα πολλά σημαντικά θέματα τα οποία πιστεύω ότι θα αξιοποιήσουμε και ως Προεδρία. Θέλω να μπω τώρα συγκεκριμένα και να προσπαθήσω να απαντήσω σε όλους τους συναδέλφους. Θα τα πάρω με τη σειρά στο θέμα της δίκαιης κατανομής των βαρών για το θέμα της μετανάστευσης. Ο ρόλος Προεδρίας είναι ουσιαστικά να διευκολύνει στην εξέβρεση κοινών τόπων σε αυτό το πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στο Ευρωκοινοβούλιο που να μην γνωρίζει τις ελληνικές θέσεις. Αυτές είναι πάρα πολύ γνωστές και έχουν κατ' επανάληψη και έχουμε κατ' επανάληψη τοποθετηθεί όλοι οι αρμόδιοι οι οποίοι βρίσκονται κοντά σας. Και πιστεύω ότι και πολλές χώρες σχεδόν όλες τις συμμερίζονται και κυρίως οι χώρες που δέχονται τον κύριο όγκο της παράνομης ε, μετανάστευσης. Υπάρχουν βέβαια και χώρες οι οποίες διαφωνούν με την πρακτική εφαρμογής κάποιων ε, κανόνων δίκαιης κατανομής βαρών. Εδώ, σε αυτό το σημείο, εγώ θα ήθελα να σας πω, να σας θυμίσω τα νούμερα τα οποία είπαμε. Είναι ουσιαστικά ένας αριθμός πάνω από το 10% του πληθυσμού. Δεν ξέρω ποια χώρα θα το άντεχε, ακόμα και αν δεν είχε οικονομική κρίση. Αυτό που έχω εγώ να πω πάντως ως ελληνική προεδρία θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε για να εξηγήσουμε το πρόβλημα και πιστεύω ότι θα βρούμε κατανόηση. Όλα αυτά έχοντας πάντα κατά νου τον ιδιαίτερο ρόλο, και αυτό το καταλαβαίνετε όλοι, που έχει μια χώρα όταν ασκεί την Προεδρία. Επαναλαμβάνω όμως, οι θέσεις μας είναι γνωστές σε όλους. Τώρα, Όσον αφορά τα, ε, τα θέματα τα οποία έβαλε, θέλω να ευχαριστήσω τον Βρετανό συνάδελφο για τα καλά του λόγια. Ε, νομίζω το τόνισα και εγώ ότι το θέμα της ε, ανάπτυξης, αν θέλετε, είναι το καλύτερο εργαλείο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ακρές πολιτικές συμπεριφορές. Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που έχει πρόβλημα παρουσίας ακραίων πολιτικών συμπεριφορών. Επίσης θα ήταν άδικο να μιλήσουμε ότι αυτό αφορά τον Ευρωπαϊκό Νότο. Τέτοια φαινόμενα υπάρχουν παντού. Και βέβαια το πρόβλημα, θα συμφωνήσω μαζί του, το πρόβλημα δεν είναι τεχνικό. Και κάτι άλλο αναφέρθηκε στο ότι δεν είναι κομματικά τα ζητήματα και βέβαια δεν είναι κομματικά. Αυτά τα ζητήματα δεν έχουν να κάνουν με κομματικές θέσεις. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι η Νέα Δημοκρατία, ένα από τα δύο κόμματα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ε, εξουσία, να το θυμίσω ότι την περίοδο που ήταν αντιπολίτευση στήριξε το 50% των νομοθετημάτων τα οποία ήρθαν στην Ελληνική Βουλή και αφορούσαν διαρθρωτικές αλλαγές. Μάλλον το 50% των νομοθετημάτων που συνολικά ήρθαν και αυτό το 50% το οποίο στηρίξαμε ήταν όλα διαρθρωτικές αλλαγές. Τώρα, ε, ακούστηκε για το θέμα της ε, χρυσή Αυγής ε, και χαίρομαι που ε, η συνάδελφος αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουμε κάνει. Ξαναείπα, το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό. Αναφέρθηκε το θέμα του παραβόλου. Αυτό δηλαδή τα 100 ευρώ που αναφέρθηκαν, το οποίο ε, λείπει ο Υπουργός Δικαιοσύνη, δεν θα ήθελα να μπω στα χωράφια του, θα ήθελα όμως να μην το αφήσουμε αναπάντητο εδώ, εάν κάποιος υποστεί βία, δεν περιμένουμε το παράβολο. Υπάρχει αυτεπάγγελτη παρέμβαση της δικαιοσύνης. Υπάρχει αυτεπάγγελτη παρέμβαση της δικαιοσύνης, άρα δεν είναι οικονομικό το ζήτημα. Ούτε δεν διαχωρίζουμε στις περιπτώσεις αυτές παράνομο και νόμιμο μετανάστη. Έτσι, εάν ο νόμιμος μετανάστης είναι αυτός που έχει υποστεί κάποιο, κάποια βίαιη συμπεριφορά, να μην τολμά να εμφανιστεί στην δικαιοσύνη. Ειδικά για αυτούς οι οποίοι έχουν υποστεί επίθεση και είναι παράνομοι μετανάστες, τους δίνεται ειδική άδεια και παραμένουν στη χώρα και για να καταθέσουν και επίσης προστατεύονται από την ελληνική πολιτεία. Και βέβαια, ε, για το θέμα του νομοσχεδίου που βρίσκεται στην ε, Βουλή για τον ε, ρατσισμό, στον κώδικα για τη μετανάστευση υπάρχει ειδική διάταξη για τα θύματα της ρατσιστικής βίας που εάν είναι παράνομοι έχουν την ίδια ευνοϊκή αντιμετώπιση με τα θύματα του τράφικη. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Τουρκίας που ρωτήσατε, έχουμε υπογράψει συμφωνία για την επιστροφή παράνομων μεταναστών από το 2001. Πρέπει να πούμε όμως ότι πρακτικά έχει εφαρμοστεί ελάχιστες φορές. Στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του Δεκεμβρίου του 2013 συνδέεται το θέμα των θεωρήσεων για Τούρκους με την εφαρμογή των επιστροφών παράνομων μεταναστών. Εμείς ως χώρα καλωσορίζουμε τη σχετική συμφωνία και περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή της. Αν αυτό εφαρμοστεί σωστά, τότε θα δούμε και το θέμα των θεωρήσεων συνολικά. Ε, Τώρα, ακούστηκε κάτι και για τα θέματα της δικαιοσύνης, πώς αντιμετωπίζει τους βουλευτές οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Θέλω να πω ότι καταρχήν, το ξαναείπαμε, ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Και αυτό δεν είναι στα λόγια, αυτό δεν είναι στα λόγια. Όποιος έχει παρακολουθήσει την υπόθεση θα δει ότι με βάση το κατηγορητήριο άλλοι έχουν προφυλακιστεί, ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής και σημαντικά, σημαντικά τη στελέχη, άλλοι έχουν, δεν έχουν μεν προφυλακιστεί, έτσι, είναι υπό περιοριστικούς όρους, άρα η δικαιοσύνη κάνει την δουλειά της ανεξάρτητα από την εκτελεστική εξουσία. Και βέβαια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε την κρίση της για να καταλήξουμε ε, στο θέμα αυτό. Επειδή ακούστηκε και η συζήτηση για τη βία, Θέλω να πω ότι η βία και ο εξτρεμισμός δεν πρέπει κανείς να τον διαχωρίζει με χρώματα. Και στην καταδίκη της θα πρέπει να είμαστε κάθετοι, και απόλυτοι. Χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Κάθετοι και απόλυτοι στην καταδίκη της τρομοκρατίας, του εξτρεμισμού και των ακραίων πολιτικών συμπεριφορών από όπου και αν προέρχεται. Τώρα, όσον αφορά για το θέμα που αναφέρθηκε για το αν υπάρχει κάποιος δρόμος για κάποιον παράνομο για να νομιμοποιηθεί. Βεβαίως υπάρχει. Εξετάζεται αναπερίπτωση κατά πόσον κάποιος παράνομος έχει καταρχήν ας πούμε αποκτήσει δεσμούς με τη χώρα. Εκείνο στο οποίο εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι είναι στις μαζικές νομιμοποίησεις. Όσον αφορά, επειδή αναφέρθηκε το θέμα των σύρων, από το 2011 μέχρι σήμερα μένουν στην Ελλάδα νόμιμα από το 2011 μένουν νόμιμα 11.300 πρόσφυγες από τη Συρία. Προσέξτε, δεν έχουν ζητήσει άσυλο. Εμείς όμως τους επιτρέπουμε να μένουν στην Ελλάδα μέχρι να τελειώσει η κρίση στην ε, πατρίδα τους. Όσον αφορά το θέμα το άλλο που αναφέρθηκε για τα στοιχεία ότι οι μετανάστες συνεισφέρουν στο 1% του ΕΠ, ε, προσωπικά θα με συγχωρέσετε δεν τη γνωρίζω αυτή τη στατιστική. Αυτό που γνωρίζω πάντως είναι ότι υπάρχει μεγάλη εκμετάλλευση όχι μόνο στην Ελλάδα όλων των παράνομων μεταναστών έτσι, Υπάρχει μεγάλη εκμετάλλευση και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε το θέμα συνολικά. Αντί να ερχόμαστε να θεραπεύουμε, θα πρέπει να πάμε στην πηγή του προβλήματος. Και θα πρέπει να πάμε στις χώρες από όπου ξεκινούν οι μεταναστευτικές ροές. Και με μία βαθμιαία προσέγγιση με τις χώρες αυτές, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να μην υπάρχει ανάγκη να φύγουν από τις χώρες τους για να έρθουν σε εμά. Δεν μιλάμε βέβαια για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει πόλεμος, εμφύλιος, ή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα γιατί έχουμε και αυτή την πραγματικότητα να μην υφίστανται για κάποιες χώρες κρατικές δομές. Εκεί λοιπόν θα πρέπει η Ευρώπη να προστρέξει και βαθμιαία ανάλογα με την πρόοδο που έχει αυτή η χώρα να βοηθάμε έτσι ώστε να μπορούμε να κλείσουμε επιτέλους αυτή τη ροή αντιμετωπίζοντας αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους που διακινδυνεύουν τη ζωή τους και γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους επιτίδιους να μπορούν να μείνουν στη χώρα τους και να προκόψουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. We have exhausted the excuse me, αν θα μπορούσαμε να αποχωρήσουμε γιατί υπάρχουν κάποιες συναντήσεις που πρέπει να κάνουμε με μέλη του Κοινοβουλίου, το οποίο δεν θα ήθελα να... για το θέμα των δύο οδηγιών Θυμόσαστε ότι στον περασμένο μα ταξίδι είχαμε συζητήσει και μαζί όταν είχατε, τη, είχατε κάνει τιμή να με επισκεφτείτε για τα θέματα των δύο οδηγιών. Okay, yeah, we... Το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να δοθούν όμω κάποιε απαντήσει από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Γεωργιάδη για να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις. Εσάς σας ευχαριστούμε. Συναδέλφους, να είσαστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Let me tell you, sure, on behalf of the Libe Committee. Εκ μέρους της Επιτροπής LIBE. θα θέλαμε να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. ταυτιζόμαστε, κατανοούμε τη θέση σας, ε, καταλαβαίνουμε τη δοκιμασία του ελληνικού λαού που μας την εξηγήσατε τόσο ζωντανά, με τόσο πάθος, καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε για να ασκήσετε την Προεδρία σας σούσεις της χειρότερης ε, κρίσης στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, σας ευχόμαστε καλή τύχη. Σας ευχόμαστε ιδιαίτερα καλή επιτυχία στα θέματά σας και στα θέματα που είναι αρμοδιότητα τη ε, Επιτροπή ΛΥΠΕ. Κυρίω για το θέμα προστασία των δεδομένων. Σα ευχαριστούμε για την συνεργασία και ακούμε τον κύριο Γεωργιάδη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα κοιτάξω να είμαι πάρα πολύ σύντομο, όσο σύντομο μπορώ, εν πάση περιπτώσει, έτσι ώστε να μην περάσω κατά πολύ το όριο των 5 και 30 που θέσατε και το οποίο έχει φτάσει ήδη. Ε, Περισσότερο ελληνοκεντρικά ήταν τα ζητήματα τα οποία ετέθησαν. Αυτό απεκόμισα ε, από, τους, ε, από τις κυρίες και τους κυρίους ευρωβουλευτές και άρα είμαι υποχρεωμένος <clears throat> ε, σε αυτό το πλαίσιο να κινηθώ. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε ε, είναι τι σημαίνει ξένος Δίας. Δηλαδή να κάνω πρώτα ένα κύκλο ε, γύρω από τα αστυνομικά ζητήματα τα οποία τέθησαν. Ξεκινήσαμε την επιχείρηση αυτή το καλοκαίρι του 2012 και ονομάσαμε ε, την επιχείρηση αυτή Ξένιος Δίας έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα τραγικά προβλήματα τα οποία υπήρχαν στα κέντρα των πόλεων μας και κατά κύριο λόγο στο κέντρο της Αθήνας. Στην προσπάθεια αυτή ε, ετέθη ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής αστυνομίας για την εξυπηρέτηση του σκοπού και πάρα πολύ γρήγορα προσπαθήσαμε να κατασκευάσουμε προαναχωρησιακά κέντρα για τους, παράνομους, για τους παράνομους μετανάστες, για τους ανθρώπους δηλαδή εκείνους που κατ' ουδέναν τρόπο δεν ε, είχαν την δυνατότητα ε, κάποιου είδου Φυσικά, στην προσπάθεια αυτή, ε, για να βρεις τους παράνομους μετανάστες, ε, ο μοναδικός τρόπος να το κάνεις είναι να τους σταματήσεις στο δρόμο και να ζητήσεις τα χαρτιά τους. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για να βρεις ε, αν κάποιος είναι παράνομος ή νόμιμος. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι έχει να κάνει αυτό σε σχέση με αυτό που ακούστηκε για τις βάσιμες υποψίες ότι ε, σταματάει η αστυνομία ε, μετανάστες στο δρόμο. Το δεύτερο ε, στοιχείο που ήθελα να αναφέρω σε σχέση με την επιχείρηση Ξένιος Δίας έχει να κάνει με τις συνθήκες κράτησης. Κανείς δεν θα υποστηρίξει ότι οι συνθήκες κράτησης σε οποιαδήποτε κέντρα, είτε προαναχωρησιακά λέγονται αυτά, ε, αλλά γενικότερα σε οποιαδήποτε κλειστού τύπου κέντρα, κανείς δεν θα υποστηρίξει ότι οι συνθήκες είναι τέλειες. Ε, θέλω να πιστεύω ότι πουθενά στον κόσμο ε, δεν υπάρχει αντίστοιχο ε, φαινόμενο παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών αλλά παροχής ανθρωπίνων υπηρεσιών. Η Ελλάδα εκείνο το οποίο έκανε είναι να ιδρύσει συγκεκριμένα προαναχωρησιακά κέντρα για τους ε, παράνομους μετανάστες, δίδοντας πρώτα απ' όλα τις σχολές της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή εκεί όπου μέχρι πρότινος ε, εσυτίζοντο και εκοιμώντο οι δόκιμοι αστυνομικοί, σε αυτούς τους χώρους ε, βρίσκονται σήμερα κατά κύριο λόγο οι, οι μετανάστες για τους οποίους μιλάμε. Άρα λοιπόν ε, σε σχέση με την ποιότητα ε, της φιλοξενίας θα μπορούσε κανείς να πει ότι από την δική μας πλευρά ε, και με δεδομένες οικονομικές συνθήκες κάναμε ό,τι καλύτερο ε, υπήρχε με δεδομένο μάλιστα ότι τα προαναχωρησιακά αυτά κέντρα δεν χρηματοδοτούνται από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια δραχμή. Σε σχέση τώρα με, την, ε, με τα φαινόμενα ρατσιστικής βίας ε, στον χώρο των ενστόλων, στον χώρο των αστυνομικών και σε σχέση με το φαινόμενο που υπόθηκε ότι ξυπνήσαμε αφού έγινε η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πολύ πριν ε, συμβεί η δολοφονία του Παύλου Φίσα, μέσα στην ελληνική αστυνομία ιδρύσαμε συγκεκριμένα τμήματα και γραφεία για την εξέταση των περιπτώσεων αντιρατσιστικής βίας. Είναι συγκροτημένα ε, πλέον δύο τμήματα και πάνω από 60 γραφεία για την αντιμετώπιση της ε, ρατσιστικής βίας στην ελληνική αστυνομία και παράλληλα για την εξέταση όλων των υποθέσεων των ε, επίορκων αστυνομικών στην ελληνική αστυνομία λειτουργεί περίφημα η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και οφείλω να ομολογήσω μπροστά σας ότι η ελληνική αστυνομία διαθέτει έναν από τους ελάχιστους φορείς εσωτερικής αυτοκάθαρσης ως οργανισμός σε σχέση με ό,τι συμβαίνει ε, ε, στην, σε υπόλοιπους φορείς στην Ελλάδα. Τώρα, ε, πολύ πιο σύντομα, ε, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Ε, εμείς εκείνο το οποίο επιδιώκουμε είναι να προχωρήσει η πρακτική εφαρμογή αυτού που ονομάζουμε ενιαίος τρόπος παροχής ασύλου στην Ευρώπη. παράλληλα, ε, σε σχέση με, την, ε, με τη στήριξη και το τι προβλέπει η ελληνική προεδρία να κάνει ε, σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που παρατηρούμε ότι σε πολλές χώρες αμφισβητούνται, εγώ ήθελα να επενθυμίσω ότι η Ελλάδα είναι το δέκατο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρείται ίσως από τα πιο παλιά μέλη πλέον και θέλω να διαβεβαιώσω ότι ως ελληνική προεδρία θα κάνουμε ε, οτιδήποτε ε, περνάει από το χέρι μας ούτως ώστε αυτοί οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να ενισχυθούν, ε, να θωρακιστούν και να εξελιχθούν εποφελία της Ευρώπης και των λαών της. Τέλος, ετέθηκε το θέμα ε, της αλληλεγγύης των κρατών. Ξέρετε, ως ε, Προεδρία η εκείνο που θα κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε τους ήδη ψηφιστέντες κανονισμούς αν και ε, επί παραδείγματι στον, στη νέα τροπολογία του κανονισμού Δουβλίνου εμείς ως χώρα είχαμε διαφωνήσει και δεν ψηφίσαμε αυτή την τροπολογία. Από την άλλη μεριά ε, σταθερή επιδίωξή μας είναι να καλλιεργηθεί, να διευρυνθεί, να μορφοποιηθεί ε, ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και αυτό θα προσπαθήσουμε ε, συνενώνοντας τις απόψεις των κρατών μελών και συνεργαζόμενοι μαζί σας και με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε οι κατευθυντήριες γραμμές που θα βγουν τον Ιούνιο που όλοι ελπίζουμε να, να, να, να τελειώσουν τον Ιούνιο ε, να εμπεριέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ε, διεύρυνση αυτής της λέξης που ονομάζουμε ε, αλληλεγγύη. Πόσο κοστίζουν τα έξυπνα σύνορα ρωτήσατε. Οφείλουμε να, οφείλω να σας πω ότι το κόστος είναι ιδιαίτερο υψηλό. δεν μπορεί να υπολογιστεί, αλλά το, στο MMF προβλέπονται περίπου 950 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κοντά στο 1 δισεκατομμύριο. Ε, σε σχέση με το Transparency Regulation, η διαπραγμάτευση ε, είναι εξαιρετικά δύσκολη και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, ε, αλλά πάντως η Προεδρία δεν μπορεί να πάει πέρα από τα, ε, από τα κράτη-μέλη σε σχέση με τα θαλάσσια σύνορα είπα και ε, στην, εισαγωγική μου ομιλία ότι ήδη έχουμε αρχίσει τους τριλόγους, τον τρίλογο ε, ελπίζουμε ότι ε, θα πάμε καλά. Τέλος, σε σχέση με θα μου επιτρέψετε μία φρασούλα μόνο σε σχέση με την άκρα δεξιά και τη Χρυσή Αυγή η, η Ελλάδα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενισχύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς και σε κάθε περίπτωση δεν θα επιτρέψει ούτε ε, στο εσωτερικό της, ούτε στους χώρους ε, της γέννησης της δημοκρατίας, δεν θα επιτρέψει να καλλιεργηθούν ε, τέτοιου είδους φαινόμενα, τα οποία άλλωστε ε, δεν τα είχαμε ποτέ στη δική μας χώρα από την ίδρυση της ως ελληνικό κράτος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Thank you for that. Thank you. Again. Σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή την ε, πολύ περιστατωμένη συζήτηση και δεν μπορώ παρά να ευχηθώ ε, και να σας καλή επιτυχία και να σας διαβεβαιώσω για τη συνεργασία με την δική μας Επιτροπή τουλάχιστον, ώστε η δική σας θητεία να, είναι, ε, να γίνει υπό τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, ιδιαίτερα για τον ελληνικό λαό, όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ε, τι περνά και πόση αντοχή έχει δείξει μέχρι στιγμή ο ελληνικός λαός για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης και τη διαχείρισή της που μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει όπως θα έπρεπε. Κυρίως λοιπόν για τους, ε, για τους Έλληνες ε, το έχουμε στο μυαλό μας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην, Ευρωπαϊκή, στην Ελληνική Προεδρία και στον ελληνικό λαό. Και αμέσως συνεχίζουμε, περνάμε στα επόμενα σημεία που έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Ας κρατήσουμε το ρυθμό, ας μείνουμε σε κίνηση διότι... Μέχρι τις 6.30 πρέπει να τελειώσουμε και έχουμε ένα-δυο σημεία να συζητήσουμε. Καταρχήν έχουμε μια κοινή συζήτηση σε σχέση με τις ε, ρυθμίσεις με την ε, Ελβετική ε, Συνομοσπονδία για το υπηρεσία στήριξης ασύλου, Λιχτενστάιν και Ισλανδία πάλι για το άσυλο. Έχουμε λοιπόν τον εκπρόσωπο εδώ της Επιτροπής για μια πολύ πολύ πολύ σύντομη παρουσίαση των ρυθμίσεων με αυτές τις χώρες για τη συμμετοχή τους στο ΙΑΣΟ, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Στήριξης Ασύλου. Σύντομα μετά τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις παρατηρήσεις τους. Εκπρόσωπος της Επιτροπής είναι ο κ. Βαντεπίερ, αν δεν κάνω λάθος. Βαντεπίερ. Ο, ο κύριος Ελ, μάλιστα. Παρακαλώ σύντομα. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο. Ο κανονισμό ΑΣΟ ε, μεριμνά για να συμμετέχουν οι Ελβετία, η Λιχτεστάιν, η Ισλανδία και η Νορβηγία ω παρατηρητέ. Αυτό το άνοιγμα στι συνδεδεμένε χώρε δεν είναι μόνο ένα λογικό βήμα που ακολουθεί την ε, σύνδεσή του στο σύστημα του Δουβλίνου, αλλά έχει και προστιθέμενη αξία της ε, χρήσης ε, των γραφείων ΕΑΣΟ, όπως είναι η ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών και προγνωμοσύνης, αλλά και έγκυρη προειδοποίηση και σύστημα ετοιμότητας. Σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών επί τη βάση του άρθρου 218 της συνθήκης, αυτές οι κοινέ προτάσεις είναι το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων με τις συνδεδεμένες χώρες. Έχουμε φτάσει σε συμφωνία μαζί τους και το τελικό κείμενο του σχεδίου ρύθμισης ε, εκπονήθηκε τον Ιούνιο του 2013. Επίσημη πρόταση επιτροπής που σας έχει υποβληθεί εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2013. Εν γέννη, οι ε, ε, λειτουργικές ρυθμίσεις θα επιτρέψουν στις συνδεδεμένες χώρες να συμμετέχουν στις εργασίες στο ΕΑΣΟ και να λαμβάνουν και να στέλνουν ε, προτάσεις για δράση στην ΕΑΣΟ. Λόγω έλλειψης χρόνου θα σας πω ποιες είναι οι βασικές ρυθμίσεις. Προβλέπεται η πλήρη συμμετοχή των συνδεδεμένων χωρών στι δραστηριότητε του Γραφείου Στήριξης, η συμμετοχή των ίδιων χωρών στον τομέα, του, στο, μάλλον στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου, οικονομική συμβολή των συνδεδεμένων χωρών στον προπολογισμό του οργανισμού θα υπολογιστεί έτσι ώστε κάθε μία συνδεδεμένη χώρα να συμβάλλει με ένα ετήσιο ποσό που υπολογίζεται σε, συμφωνία με το, ε, σε σχέση με το ΑΕΠ για όλα τα συμμετέχοντα κράτη και έχουμε επίσης τη δυνατότητα να έχουμε μια επιπλέον συμβολή των συνδεμένων χωρών σε περίπτωση κρίσης. Επιπλέον, η συμφωνία προβλέπει ε, μετά από αίτημα των συνδεμένων χωρών την δημιουργία μιας επιτροπής που αποτελείται από εκπροσώπους ε, της Επιτροπής και των συνδεμένων χωρών, δεν έχει αρμοδιότητα λήψη απόφασης και παρακολουθεί τη σωστή ε, εφαρμογή των ρυθμίσεων και αυτός και εξασφαλίζει τη συνεχιζόμενη ροή πληροφοριών. Ε, τέλος, εμείς στην Κομισιόν θεωρούμε πως ε, το σχέδιο ρύθμισης που έχετε εδώ καλύπτει τα σχετικά με τον κανονισμό και γι' αυτό θα πρέπει να είναι αποδεκτό για την Ένωση. Και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή, τον κύριο Και τον ευχαριστώ κιόλας επειδή έλαβε υπόψη του τον ε, περιορισμένο χρόνο που έχουμε. Θα ήθελε η Προεδρία να πει κάτι γι' αυτό πρώτο προχωρήσουμε στους ευρωβουλευτές. Παρακαλώ. Πόσο. Okay. You go ahead. Ονομάζομαι Μάλιος κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για το λόγο. Να ήθελα να προσθέσω πολύ σύντομα κάτι σε αυτά που μόλις ε, δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί ο φάκελος αυτός. Ήδη σχεδιάζουμε στις 28 Ιανουαρίου, την επόμενη εβδομάδα, ένα Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, όπου θα συζητήσουμε την πρόταση της Επιτροπής και βασισμένη στα αποτελέσματα της συζήτησης αυτής και χωρίς να θέλουμε να προδικάσουμε το αποτέλεσμά της. Υποθέτουμε ότι το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνουν το κείμενο. Σχεδιάζουμε λοιπόν να το υποβάλουμε στους γλωσσομαθείς νομικούς και έπειτα να το υποβάλουμε για έγκριση στην Κορεπέρ και το Συμβούλιο. Ελπίζουμε μέσα στο Φεβρουάριο, το συντομότερο όπως και να έχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μετσόλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομη. θα είμαι επικεφαλής για το φάκελο αυτό και είναι και τιμή μου γιατί είναι η πρώτη έκθεση που αναλαμβάνω σε αυτήν την Επιτροπή. Συμφωνώ με τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει η πολιτική αυτή που είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να επιτύχουμε τους στόχους μας. Η συμμετοχή αυτών των συνδεδεμένων χωρών θα προσθέσει μια πολύ σημαντική διάσταση στην ΕΙΑΣΟ και θα διευκολύνει και την ε, ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα χαρώ πάρα πολύ να ασχοληθώ με την έκθεση αυτή και να συναντηθώ με τους εκπρόσωπους των άλλων πολιτικών ομάδων και ελπίζω να οδηγηθούμε γρήγορα σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν πολύ σύντομοι. Ακούσαμε λοιπόν την εισηγήτρια θα ήθελε κάποιος από τους κοιόδης εισηγητέ που βρίσκεται στην αίθουσα να σχολιάσει. Όχι. Εφόσον όχι, θα ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Για όλες αυτές τις συμφωνίες, τις ρυθμίσεις με τις ε, χώρες ε, και τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το άσυλο. Τελείωσαμε λοιπόν και έχουμε ένα τελευταίο σημείο να εξετάσουμε τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας για την επανειστοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια. Θα ακούσουμε τώρα την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον κύριο Τούντοράτσε για τις ε, νεότερες εξελίξεις σχετικά με την Συμφωνία Επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας στις 16 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους υπεγράφει αυτή η συμφωνία στην Άγκυρα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από ψηφοφορία. Ωστόσο, πριν ψηφίσουμε, στις 6-7 Μαΐου δηλαδή, έχουμε καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει για τις νεότερες εξελίξεις. Θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Τοντοράτζε, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βρίσκεται στην αίθουσα. Ε, κύριε Πρόεδρε, μόλις τώρα έρχεται. Θα είναι εδώ σε λίγο. Ωραία, θα περιμένουμε τότε και ας διακόψουμε για ένα λεπτό και μετά θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Let's move on. Mr. Κύριε Τούτου, εκπρόσωπο τη ε, Επιτροπή, καλώ ήρθατε. Θα μα μιλήσετε για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία για την επανειστοχή προσώπων. Θα ήθελα να κάνω την παρουσίασή σα, ούτω ώστε να δώσω το λόγο στον εισηγητή και συνεχεία στου ευρωβουλευτέ. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που με περιμένατε. Θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κύριου Μασερβίση που ήθελε να έρθει εδώ, γιατί η Τουρκία είναι πολύ σημαντικός φάκελος για τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και θα ήθελε ο ίδιος να σας κάνει την παρουσίαση, αλλά για λόγους που γνωρίζετε φαντάζομαι και για, λόγω εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σήμερα δεν μπόρεσε να έρθει τελικά. Ούτως ή άλλως, η υπογραφή της συμφωνίας ήταν ε, μια πολύ σημαντική πολιτική στιγμή στη σχέση μας με την Τουρκία. Ξέρετε ότι η τελευταία ενημέρωση που κάναμε στην Επιτροπή ήταν το Μάιο του 2013 και το Μάιο δεν ε, μπορούσαμε να σας πούμε ότι είχε σημειωθεί μεγάλη πρόοδο στις συζητήσεις μας με τους Τούρκους εταίρους γιατί για τη Συμφωνία Επανειστοχής δεν υπήρχε καμία απολύτως κίνηση. Τι προκάλεσε την αλλαγή, μπορεί να ρωτήσει κάποιος. Η προσφορά που κάναμε για τις θεωρήσεις ήταν πολύ σημαντική για τους Τούρκους. Παρενθετικά να πω εδώ ότι αυτό είναι ένα θετικό αποτέλεσμα της ε, συνολικής προσέγγισης που έχουμε στη μετανάστευση και την κινητικότητα, που εδώ και χρόνια προωθούμε και που τώρα δίνει καρπούς. Όχι μόνο στη Νότια Μεσόγειο, αλλά και στην περίπτωση της Τουρκίας τώρα πια. Με αυτή την προσφορά λοιπόν επιτάπητος, τελικά είχαμε αυτή την κίνηση από πλευράς Τούρκων. Κάνα αυτή την πρόοδο και έδειξαν ανοιχτό πνεύμα το Δεκέμβριο για να υπογράψουν τη συμφωνία. Τώρα, τι υπάρχει σε αυτή τη συμφωνία, τι εμπεριέχεται στο κείμενο. Το πρώτο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι είναι μια κλασική συμφωνία που η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει γενικά με τρίτε χώρε, δηλαδή ω προ το περιεχόμενο, ω προ τι διατάξει, ω προ εγγυήσει. Μοιάζει πάρα πολύ με τα όσα έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια σε όλε τι συμφωνίε επανεισδοχή. Σε ποιον απευθύνεται τώρα. Έχουμε την ε, κλασική μεταβλητή γεωμετρία. Δανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο. Τίποτα άλλο όμω, καμία άλλη εξαίρεση, ισχύει για όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καλή η συμφωνία και ω προ το περιεχόμενο, γιατί όχι μόνο καλύπτει διατάξει που αφορούν την ε, επανεισδοχή Τούρκων υπηκών, μεταπών δηλαδή, αλλά και υπηκόσου των χωρών που έχουν ε, μπει στην ε, Ευρωπαϊκή Επικράτεια μέσω Τουρκία. Δεν χρειάζεται να σα εξηγήσω εδώ πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί η Τουρκία εκπροσωπεί αυτό που εκπροσωπεί στι μεταναστευτικέ ροέ προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα δικαιώματα και τι εγγύησει, όπω σα είπα, είναι κλασικό, συνηθισμένο κείμενο. Επομένω, έχει όλε τι διατάξει και προβλέπει όλε τι εγγύησει, διεθνή προστασία, δικαιώματα, ασφαλιστικέ δικλείδε που περιμένει οποιοδήποτε και που ισχύουν στη διαδικασία επανεισδοχή. Όλα αυτά θα ισχύσουν υπό τη συμφωνία. Για την εφαρμογή τώρα. Για τέτοιε συμφωνίε επανεισδοχή παρακολουθούμε πάντα εκ του τη διαδικασία. Θα υπάρξει μια κοινή επιτροπή επανεισδοχή όπου η Κομισιόν, η Τουρκία αλλά και οι αρμόδιες αρχές θα συνεδριάσουν για να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Για να ολοκληρώσω και να αφήσω και χρόνο για τις ερωτήσεις και απαντήσεις είναι μια πολύ θετική στιγμή αυτή. Νομίζουμε ότι είναι μια ιστορική στιγμή στις σχέσεις μας με την Τουρκία και δείχνει επίσης και την κατάσταση στην οποία έχει φτάσει ο πολιτικός διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Είναι ισορροπημένο το κείμενο. Πιστεύουμε ότι θα, έχουμε, ότι θα υπάρχει θετική επίπτωση από αυτό το κείμενο στην μείωση της ε, παράτυπης μετανάστευσης. Γιατί πιστεύουμε ότι πραγματικά είναι εφαλτήριο η ενδιάμεσο σταθμό η Τουρκία για τη μετανάστευση. Η κυρία Σόμερ θα μας κάνει τώρα την παρουσίασή της, είναι Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα, στις 16 Δεκεμβρίου λοιπόν του 2013 υπεγράφει συμφωνία επανειστοχής στην Άγκυρα μετά από πάρα πολλέ καθυστερήσεις από εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω ήδη αναφέρθηκε και χωρίς ε, όμως ε, να μην υπάρχουν και απαιτήσει από την πλευρά της Τουρκίας. Ε, δηλαδή, ταυτόχρονα με την υπογραφή της συμφωνίας να εισέλθει σε διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις ε, διευκολύνσεις έκδοσης θεώρησης για Τούρκους υπηκόους από την ευρωπαϊκή πλευρά. Αυτό υπεγραφή άνοιξε μάλλον ταυτόχρονα με την υπογραφή της Συμφωνίας 16 Δεκεμβρίου. Ε, η συμφωνία αυτή θα συνεισφέρει πολύ στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τουρκία και θα είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμη για την καταπολέμηση της διασωνοριακής εγκληματικότητας, ιδιαίτερα του εμπορίου και της διακίνησης ανθρώπων. Όχι μόνο όμως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που θα υποφεληθεί από τη συμφωνία αυτή, αλλά και η Τουρκία, διότι η Τουρκία πλέον έχει προοπτική για διευκόλυνση και απελευθέρωση το, της έκδοση έκδοσης ε, θεωρήσεων και επίσης ε, τεχνική συνεργασία όσον αφορά την φύλαξη των συνόρων. Η Υπήρξαν όμως ορισμένες ε, επικρίσεις σχετικά με τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου. Δεν ήταν ε, όλα τα κράτη-μέλη σύμφωνα με αυτήν την ε, απελευθερώση, αυτή τη διευκόλυνση θεωρήσεων και από την άλλη ούτε η Τουρκία τήρησε τις υποσχέσεις της. Μέχρι τώρα έχει απλώς μονογραφήσει την συμφωνία και δεν έχει τηρήσει καμία σχεδόν υποχρέωση. Για παράδειγμα, δεν αποδέχεται την ακαιρεότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό φαίνεται και από την αρνητική της στάση έναντι της Κυπριακής Προεδρίας το 2012. Επίσης ε, ε, διαπιστώνονται παραβιάσεις ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, παραβίαση της ελευθερίας του τύπου και πάρα πολλά άλλα σημεία στα οποία η Τουρκία έχει οπισθοχωρήσει και δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο. Ο μαζικός αυτός περιορισμός και παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών αντιβαίνει στα πολιτικά κριτήρια της Κοπενχάγης για την προταξιακή διαδικασία που πρέπει να πληρεί η Τουρκία έτσι ώστε να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τις θεωρήσεις. Ωστόσο, να τονίσω ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τις θεωρήσεις Χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται διάλογος και εδώ να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει και να εισέλθει στο, στο διάλογο αυτό ενωμένο. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την κυπριακή πλευρά. Ωστόσο δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσει η Τουρκία το θέμα της Κύπρου. Εμείς πάντως σε κάθε περίπτωση ως ευρωβουλευτές θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχιστεί ο διάλογος. Η διευκόλυνση λοιπόν αυτή για τις εθεωρήσεις αφορά κυρίως σε Τούρκους υπηκός που θέλουν να ταξιδεύουν χωρίς πολλούς περιορισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο δικός χάρτης ο οποίος έχει ζητήσει η Τουρκία για ε, τη διευκόλυνση έκδοσης θεωρήσεων. Αυτό όμως θα συμβεί μόνο όταν η Τουρκία πληρεί τις προϋποθέσεις που έχουν ήδη τεθεί. Το σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα μεταξύ άλλων. Μετά την ε, κύρωση μιας τέτοιας συμφωνίας η Τουρκία θα υποφεληθεί από τεχνική και οικονομική υποστήριξη στη φύλαξη των ε, συνόρων, την εποπτεία των συνόρων και την ε, αστυνομία, την καταπολέμηση, όπως είπα, του διασυνοριακού εγκλήματος και ιδίως της διακίνησης ανθρώπων και του τράφικινγκ. Πρέπει όμως να διασφαλιστεί η τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλους, για ε, ευάλωτες ομάδες, για μετανάστες και για μειονότητες. Το αργότερο μέσα σε τρία χρόνια αναμένεται να φτάσουμε στο τελικό αυτό στάδιο για την, ε, για την έκδοση θεωρήσεων για Τούρκους ε, υπηκόους. Ωστόσο δεν πρέπει να αφήσουμε να δεχτούμε τις πιέσεις της Τουρκίας διότι πρέπει πραγματικά η Συμφωνία Επανεστοχής να κυρωθεί και να εφαρμοστεί πλήρως. Αυτό συνεπάγεται και την ε, κύρωση από το τουρκικό κοινοβούλιο. Χρειάζεται αύξηση της ασφάλειας των συνόρων με την Τουρκία και εδώ να πω ότι θα παρατηρούμε πολύ στενά τις εξελίξεις και δεν θα δεχτούμε καμία περιττέρω καθυστέρηση από πλευράς της Τουρκίας. Αυτά κύριε Πρόεδρε νολίγησε στην ε, έκθεσή μου. Ελπίζω στην στήριξή σας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Απόσκουρτ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ την υπόγραφη της Συμφωνίας Επανιστοχής τον Δεκέμβριο που μας πέρασε και την έναρξη του διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας έχουν ε, λινάσει τα τελευταία χρόνια. Και ελπίζω ότι ο διάλογος ε, αυτός να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την συνέχεια του διαλόγου. Αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ε, διαδικασία ολοκλήρωσης της Τουρκίας, τη διαδικασία ένταξης, συγγνώμη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι χρειαζόμαστε αυτή τη συμφωνία για να καταπολεμήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την μετανάστευση από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συμφωνία θα είναι ωφέλιμη για όλους. Εμείς θα παρατηρούμε στενά εξελίξεις και θα προσπαθήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσουμε την Τουρκία στην εφαρμογή της. Είναι όμως το χέρι της Τουρκίας να δεσμευτούν πλήρως για την πλήρη εφαρμογή και πλήρη λειτουργία των ε, διατάξεων. Μετά από αυτό και οι δύο πλευρές θα επωφεληθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να μην εμποδιστούν οι Τούρκοι υπήκοοι και όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της συμφωνίας αυτής είναι κάτι που είναι εξαιρετική σημασίας και επίγον για τους Τούρκους ε, πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω λάβει πάρα πολλές ε, επιστολές και μηνύματα τα ε, οποία εκφράζουν ανησυχίες για την κατάσταση των Τούρκων υπηκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί έχουν καταφύγει στην γρήγορη απέλαση Τούρκων υπηκών οι οποίοι είναι, διαμένουν προσωρινά σε κάποιο από τα κράτη-μέλη. Επίσης, έχω διατυπώσει γραπτές ερωτήσεις ε, για αυτό το θέμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η απάντηση που έλαβα επιβεβαιώνει αυτά. Η συμφωνία αυτή διευκολύνει μόνο την διαδικασία για τους ε, για όσους διαμένουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για εκείνους που έχουν διάρκεια μακράς παραμονής και για όσους ε, εισέρχονται για επανένωση με μέλη της οικογένειάς τους. Αυτά είναι σημεία που θα ήθελα βέβαια και να μάθω μερικές πληροφορίες παραπάνω. Πιστεύω πως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ασκήσει έλεγχο και να διαπιστώσει εάν όντως παραβιάζονται δικαιώματα Τούρκων πολιτών. Ελπίζω επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να ε, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της Συμφωνίας Επανιστοχής. Ε, διότι το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να πληροφορούμαστε για τα ε, προβλήματα της συμφωνίας αν αυτά υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ποσκούρτ. Σα euh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου θέλω να εκφραστώ εξ ονόματος της ομάδας και να σας πω ότι χαιρόμαστε για αυτή τη συμφωνία μετά από πολλά χρόνια διαπραγματεύσεων, ε, παύσεων ε, και ε, ξανά διαπραγματεύσεων. Είμαι ευτυχής που φτάσαμε επιτέλους σε ένα κείμενο το οποίο θα ψηφίσουμε ελπίζω αύριο. Το κείμενο αυτό βέβαια θα είχε αντίκτυπο και στη διεθνή στο διεθνές προσκήνιο, γιατί νομίζω ότι ο Πρωθυπουργό Ερντογάν συναντά, ενώ συζητάμε αυτή τη συμφωνία, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου με θέμα την πρόσφατη δικαστική μεταρρύθμιση που γίνεται στην Τουρκία και που αυτή η επικαιρότητα ταυτόχρονα έχει ε, κυλιδωθεί από σκάνδαλα διαφθοράς, ε, όσον αφορά δηλαδή την απόφαση που πήρε ο Πρωθυπουργός, ο Τούρκος Πρωθυπουργός, για, ε, για μέτρα καταστολής των αντιδράσεων. Τώρα, υπάρχουν ε, πιο συγκεκριμένε ανησυχίε, αλλά και πιο γενικότερε ανησυχίε, συγκεκριμένε ανησυχίε όσον αφορά την ε, μεταρρύθμιση την δικαστική στην Τουρκία, γιατί αυτή η δικαστική μεταρρύθμιση που γίνεται δεν ακολουθεί πραγματικά ε, το στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, φαίνεται να ενισχύει το σύστημα σε αντίθεση με τις βασικές αρχές, δηλαδή τις αρχές της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, του ελέγχου του ε, εκτελεστικού στη ε, δικαστικό μηχανισμό. Βλέπουμε δηλαδή πολύ μεγάλη διεξουσία στις αστυνομικές αρχές και στις δικαστικές αρχές από τα μέσα του Δεκεμβρίου. σε σχέση με τις ε, θεμελιώδεις αρχές, δηλαδή όσον αφορά την ε, σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, την ελευθεροτυπία και κάποια μέτρα φυλάκισης βουλευτών ή που θίγουν την ανεξιθρησκεία και που έχουν αναφερθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία εκφράζουν τις ανησυχίες τους. Ωστόσο, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας και εγώ και στηρίζω την προσέγγιση όσον αφορά την επανεισδοχή, δηλαδή τη συμφωνία επανεισδοχής και, την σύμφωνη, και, την, και, ελπίζω ότι θα εγκριθεί αύριο. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ δε το ότι έχω το λόγο για να θυμίσω ένα στοιχείο το οποίο επανέρχεται σε κάθε συζήτηση πριν την ψηφοφορία για τις συμφωνίες επανεισδοχής είναι οι γενικές επιφυλάξεις που εκφράζω κάθε φορά και που δυστυχώς δεν καταλήγουν, τουλάχιστον όχι γρήγορα, στα αυτιά της Κομισιόν όσον αφορά την αξιολόγηση και την παρακολούθηση ε, αυτών των συμφωνιών επανεισδοχής και ε, αναφέρομαι κυρίως στις διαπραγματεύσει συμφωνίας επανεισδοχής με το Πακιστάν. Δεν μας αρκεί σε εμάς τους Ευρωπαίους το να ε, το οριοθετούμε τα πράγματα μέσω συμφωνιών επανεισδοχής, θεωρήσεων και έπειτα να ανοίγουμε τα σχήρας μας. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και εδώ και πάρα πολύ καιρό πόσο μπορεί να είναι πρόσκαιρο και επικίνδυνο για ορισμένους πολίτες το να επιστρέψουν αν δεν υπάρχει στο τεχνοκρατικό ευρωπαϊκό μας ε, ε, ορολογία αυτό που λέμε επαναξελόγηση, παρακολούθηση αυτών των ανθρώπων που αποτελούν αντικείμενο μιας επανεισδοχής. Επαναλαμβάνω λοιπόν το αίτημα για ενημέρωση και αξιολόγηση των συμφωνιών επανεισδοχής των ισχυουσών ή αυτές των οποίων έχει υλοποιηθεί η εφαρμογή. Μια πραγματική λοιπόν αξιολόγηση, όχι απλά στατιστικές ε, και πληροφορίες, μια πραγματική αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρώπων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας επανεισδοχής. Θα ήθελα, υπογραμμίζοντας την ποιότητα της έκθεσης και της ε, εργασίας που έχει ήδη γίνει, λοιπόν, να θυμίσω πως ο διάλογος ο οποίος έχει εγκαθιδρυθεί ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρώπη μας ε, θα όφιλε να συνεχιστεί Και επίση να υπογραμμίσω πως είναι πολύ σημαντικό να γίνεται μια συγκεκριμένη αναφορά στην κατάσταση των προσφύγων από τη Συρία. Κύριος, που δεν θα πρέπει να ξεχαστούν ή εν πάση περιπτώσει όλοι όσοι χρήζουν διεθνούς ε, προστασίας και βρίσκονται σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Και να πω ότι για αυτούς δεν θα πρέπει η Τουρκία να εκμεταλλευτεί τη Συμφωνία Επανεισδοχής και να τους αφήσει στην άκρη, να τους ξεχάσει. Να πω τέλος ότι αυτές οι συμφωνίες είναι εξαιρετικά σημαντικές σε συνδυασμό με την απελευθέρωση ή τη διευκόλυνση των θεωρήσεων για να ανοίξει η Ευρώπη στην υποδοχή ερευνητών, φοιτητών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και να διευκολυνθούν έτσι οι επαφές ανάμεσα στους πολίτες πράγμα που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει αποτελεσματικός και συγκεκριμένος διάλογος. Ε, στον τομέα τον οικονομικό, τον πολιτιστικό, αλλά και τον ανθρωπιστικό και τον επιστημονικό. Εδώ τελειώνω, Προέδρε, και είμαι υπέρ της έκθεσης. Ευχαριστούμε, κυρία Σαργεντίνη. Παρακαλώ. Εξήμιση πρέπει να τελειώσουμε. Έχετε το υπόψη Ναι, ευχαριστώ. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Οι πράσινοι στο παρελθόν ήταν πάντοτε αντίθετοι ε, σε τέτοιες συμφωνίες επανεισδοχής. Ήμασταν ανέκαθεν κατά, διότι δεν μπορούμε να δεχτούμε να υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου των ευρωπαϊκών συνόρων και όλο αυτό το πρόβλημα της μετανάστευσης, ε, της ανεπιθύμητης μετανάστευσης, να, στην ουσία να μετεγκαθίσταται στις τρίτες χώρες. Πακιστάν, είδαμε τι έγινε, είδαμε με τη Λιβύη, με την Τινησία και για την Τουρκία το ίδιο απαράδεκτη μου φαίνεται αυτή η συμφωνία. Αύριο, στην στιγμή της ψηφοφορίας, εμείς θα προτείνουμε ένα αναλλακτικό ψήφισμα, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας κάνω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο, κυρία Μπόσκουτ. Όταν λέτε ότι πρόκειται για μια κατάσταση όπου όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Μα ποιος βγαίνει κερδισμένος. Οι μετανάστες που δεν έχουν το δικαίωμα ασύλου και τους στέλνουμε πίσω στην Τουρκία, ε, μια χώρα που δεν έχουν να κάνουν τίποτα, γιατί δεν είναι καν ε, Τούρκοι όπου δεν γίνεται δεκτή η Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και όπου οι σε άσυλο οι πρόσφυγες που έρχονται από χώρες ε, ευρωπαϊκές είναι οι μόνοι οι οποίοι γίνονται δεκτοί. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες για την υποδοχή των μεταναστών στην Τουρκία. Είτε έχουν είτε δεν έχουν χαρτιά. Και έπειτα, όταν μου λέτε ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση καλύτερη ποιότητα, φυσικά και συμφωνώ μαζί σα, θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώ τι συμβαίνει, τι γίνεται με του μετανάστε που του στέλνουμε πίσω στην Τουρκία. Αλλά πραγματικά αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Θα ξέρουμε τι γίνεται. Και άμα ξέρουμε ότι πάνε καλά τα πράγματα, θα συνεχίσουμε να του στέλνουμε πίσω. Ξέρουμε όμω πάρα πολύ καλά ότι στην Τουρκία οι εγκαταστάσεις δεν είναι στο ύψος ε, των περιστάσεων Ξέρουμε, έχουμε και το παράδειγμα των θεωρήσεων και ξέρουμε ότι με, στην ουσία μεταφέρουμε τον έλεγχο των συνόρων στην Τουρκία, στο Ιράκ, εν πάση περιπτώσει όλες αυτές τις ηλιόλουστες χώρες. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της δραστηριότητα παρακολούθησης ή ελέγχου, κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό για να τους ξαποστείλουμε στην ουσία push back Τέτοιου είδους εγγύηση δεν υπάρχει πουθενά. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, για τους ε, Τούρκους ε, υπήκοους Βεβαίω θα μπορούν να ταξιδεύουν πιο ελεύθερα. Αυτό είναι καλό, σε αυτό είμαι υπέρ, αλλά για την επανεισδοχή όχι, διαφωνώ και σίγουρα δεν είναι μια κατάσταση που όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Ο χαμένος είναι πάντα μετανάστες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Άινστ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να το διατυπώσω με προσοχή. Να πω ότι σε αυτή την κατάσταση που έχετε περιγράψει είναι πιστεύω ανεύθυνο να υπογράψουμε μια τέτοια συμφωνία. Και τι ακούσαμε, να επαναλάβω. Οπισθοχωρήσεις, ε, κατά της ε, δημοκρατίας, παραβιάσεις, κανένας επικοδομητικός διάλογος. Όλοι οι συνάδελφοι έχουν μιλήσει γι' αυτό, για παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων, για καμία πρόθεση από μέρου της Τουρκίας, ε, ιδιαίτερα στους τομείς της δικαιοσύνης να κάνουν βελτιώσεις και αυτή τη στιγμή το να εγκριθεί μια τέτοια συμφωνία είναι κάτι που εγώ το θεωρώ τουλάχιστον ανεύθυνο. Ε, δεν θέλω καν να μπω στην διαδικασία να παρομοιάσω τη συμφωνία αυτή με άλλες συμφωνίες. Και κάτι άλλο ότι φυσικά η ελευθέρωση της θεώρησης θα ήταν ένα δωράκι που θα δίναμε στην Τουρκία, χωρίς καμία ανταπόκριση, χωρίς καμία ανταπόδοση. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς, ποιον αφορά αυτή η συμφωνία. Τούρκους υπηκόους. Ποιον αφορά λοιπόν αυτή η συμφωνία, ποια είναι τα τρίτα κράτη τα οποία αναφέρεται, η Συρία, το Ιράκ, ποια άλλη. Τρίτον, ε, όσον αφορά αυτούς που αφορά η συμφωνία αυτή, ε, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Τι γίνεται με την Κύπρο, τι γίνεται με τη Βόρεια, με το Βόρειο τμήμα. Έχω βρει κάποιες πληροφορίες μετά από αναζήτηση που έκανα μόνη μου, όμως δεν με ικανοποίησαν και θα ήθελα εσείς να μου πείτε τι θα γίνει με την Κύπρο. Πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι αν τους κάνουμε ένα τέτοιο δώρο, είναι κάτι που είναι όχι μόνο τελείως ανεύθυνο, αλλά και τελείως αντίθετο στις αρχές μας. Ωστόσο, όμως, μου φαίνεται πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας. Δεν είμαι κατά της ελευθέρωσης των θεωρήσεων, όμως όχι με τέτοιες προϋποθέσεις και με τέτοιο πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπρόντς. Αναρωτιέμαι γιατί πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους οι χώρες αυτές για να πάρουν πίσω τους υπηκόους τους. Φυσικά ο καθένας έχει ένα προσωπικό δικαίωμα να επιστρέφει, να πηγαίνει όπου θέλει. Ωστόσο, στην περίπτωση ενός τα μετανάστη που επιστρέφεται χωρίς τη θέλησή του, κάπου είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Πιστεύω πως αυτή τη συμφωνία η Τουρκία θα ε, πρέπει να συμφωνήσει να πάρει πίσω τους ειδικούς της υπηκόους. Βέβαια το αν θα γίνει αυτό και πότε θα γίνει αυτό είναι άλλο θέμα και και η συγγήτρια και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι είχαν δίκιο που αναφέρθηκαν για τις αμφιβολίες τους για αυτό το σύστημα ελευθερώσης των θεωρήσεων. Διότι αυτό κινδυνεύει στο τέλος να μετατρέψει, να αλλάξει την κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ. Πρωτού επιστρέψουμε στην συγγήτρια για τα τελευταία της ε, σχόλια. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να απαντήσει στα σχόλια και τις ανησυχίες της παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών. Κύριε Τεντοράτσε. Να απαντήσω τώρα σε ερωτήσεις. Θα τις ομαδοποιήσω θεματικά. Τα προβλήματα στην Τουρκία καταρχήν. Γιατί η Κομισιόν παραβλέπει τα προβλήματα στην Τουρκία τα, προβλε... τα παραβλέπει όντως και γιατί πόσα υποβάλλεται στο τραπέζι η συμφωνία αυτή δεδομένης πολιτικής κατάστασης στην Τουρκία. Αντίθετα με κάποιες από τις απόψεις που εκφράσαν οι ευρωβουλευτές, εγώ πιστεύω ότι ο διάλογος για τις θεωρήσεις ακριβώς αυτό θέλει να κάνει. Θέλει, δηλαδή, να γίνει, να εξασφαλίσει ένα πολιτικό και τεχνικό διάλογο με τη συγκεκριμένη χώρα και προκειμένου την Τουρκία. Υπάρχουν ε, τέσσερις άξονες, 80 ορόσημα. Και κοιτάμε δηλαδή σημείο προς σημείο, ορόσημο προς, προς ορόσημο, ποια είναι η πρόοδος που έχει σημειώσει η χώρα. Ε, δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, επιδόσεις της χώρας σε κάθε ένα από αυτά τα 80 ορόσημα. Σε αυτή τη ε, διαδικασία που έχουμε θεσπίσει, το γεγονός ότι έχουμε διάλογο για τις θεωρίες με την Τουρκία, δεν θα λέγω ότι μας εξασφαλίζει κάτι, ότι είναι μια εγγύηση από μόνο του, αλλά τουλάχιστον θέτει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια θέση όπου τουλάχιστον μπορεί να συζητήσει με την Τουρκία αυτά τα σημεία και να μας δώσει πραγματικές ε, εγγυήσεις ε, για ότι κάνει σε αυτούς τους τέσσερις ε, τομείς. Πώς περνάει η νομοθεσία, πώς βελτιώνει την νομοθεσία της και μόνο όταν μας ικανοποιήσει με τις απαντήσεις, μόνο όταν μας πείσει ότι έχουν υλοποιηθεί αυτά τα ορόσημα, τότε μόνο θα σας προτείνω σε εσά και στο συνομοθέτη σας στο Συμβούλιο το να συμπεριλάβουμε την Τουρκία στον θετικό κατάλογο. Επομένως, πρόκειται για μια διαδικασία με συγκεκριμένα στοιχεία, ούτως ώστε να διασκεδαστούν οι ανησυχίε όλων. Να πιστούν ότι δεν αγνοούμε την κατάσταση στην Τουρκία, αντίθετα. Είμαστε σε επαφή με την Τουρκία, με τους σωστούς ανθρώπους και έχουμε το σωστό πλαίσιο για να συζητήσουμε τα σημαντικά αυτά σημεία. Κύπρος, άλλο σημείο. Μια άλλη ανησυχία. Και εκεί θέλουμε να είμαστε σίγουροι, δεδομένης της ιστορίας των σχέσεων της Τουρκίας με την Κύπρο. Η απόλυτη προτεραιότητά μας είναι να έχουμε μια συμφωνία επανεισδοχής χωρίς επιφυλάξεις. Και σας επιβεβαιώνω ότι η συμφωνία που έχουμε υπογράψει με την Τουρκία δεν έχει τέτοιες. Να είμαστε ξεκάθαροι στη θέση της Κομισιόν, επίσης, και για να πιστείτε θέλω να σας πω ότι μία επιστολή που συνυπογράφηκε από, την, ε, από τους επιτρόπους ε, Μάτσομ και Φούλε εστάλθη στην Τουρκία για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση της Κομισιόν σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας και τα θέματα της Κύπρου. Υπάρχει ένας σαφής μηχανισμός. Θα προσέξουμε πολύ προσεκτικά τι κάνει η Τουρκία σε σχέση με την Κύπρο και αν δούμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, τότε έχουμε το μηχανισμό για να αντιδράσουμε. Τρίτο θέμα τα δικαιώματα των Τούρκων πολιτών που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε και ο Ευρωβουλευτής, μας υποβάλλεται διάφορες γραπτές ερωτήσεις. Και ελπίζουμε ότι οι απαντήσεις που σας έχουμε δώσει γραπτός να σας διασκεδάζουν τις ανησυχίες. Αν θέλετε και άλλες διαβεβαιώσεις, μπορώ να σας πω σήμερα ότι η συμφωνία από μόνη της δεν δημιουργεί πρόβλημα στα δικαιώματα των Τούρκων πολιτών που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να υποφεληθούν από την προστασία, τα δικαιώματα, τις διαδικασίες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, εκεί όπου διαμένουν δηλαδή. Το θέμα της ε, επαναξιολόγησης της Συμφωνίας Επανεισδοχής, πολύ σημαντικό ερώτημα, μας ανησυχεί και εμάς, μας απασχόλησε πάρα πολύ. Μία θετική εξέλιξη είναι ότι απέναντι στο Πακιστάν, ας πούμε, σωστά το αναφέρατε, ως μια άλλη τρίτη χώρα όπου μια τέτοια συμφωνία επανεισδοχής υπάρχει και η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των επιστροφών είναι πολύ σημαντική και είναι σημαντικό να γίνεται. Σε αγγέλω σήμερα ότι έχουμε υπογράψει ένα πιλωτικό πρόγραμμα, τον IOM, για να εξετάσουμε την ένταξη των ατόμων που επιστρέφονται στο Πακιστάν. Ε, υπάρχουν αποτελέσματα στα πλαίσια αυτού του πιλωτικού προγράμματος Παρακολουθούμε τους ανθρώπους που επιστρέφουν στο Πακιστάν και αυτή την πρόβλεψη θα την συμπεριλάβουμε και στις συμφωνίες με άλλες τρίτες χώρες, όπου έχουμε σημαντικές επιχειρήσεις επιστροφών. Η Τουρκία, ας πούμε, είναι μια άλλη τέτοια τρίτη χώρα με την οποία ένα πρόγραμμα τέτοιου τύπου θα δημιουργηθεί. Θα παρακολουθούμε τη συμφωνία πολύ προσεκτικά και μέσω τέτοιων project θα εξετάσουμε εκ του σύνεγγυς την ένταξη των ατόμων που επιστρέφονται στις χώρες τους. Αυτά ευχαριστώ. mean, we run out of time and uh, Δεν έχουμε χρόνο. Τελευταία η συγγήτρια. Θέλουν και άλλοι όμως να πάρουν ε, το λόγο. κυρία Μποσκούρτ. Και η κυρία Έντς. Πρώτα κυρία Μποσκούρτ, αλλά σύντομα παρακαλώ. Θέλω να αντιδράσω. Πολύ σύντομα γιατί ουσιαστικά απευθυνθήκατε με ρωτήσεις σας σε αυτά που είπα εγώ. Επομένως, λογικό να αντιδράσω σε αυτά που με ρωτήσανε. Αναφέρατε κάποια από αυτά τα πράγματα που είπα, αλλά τουλάχιστον όταν παραθέτετε αυτά που λέω, να τα παραθέτετε σωστά και να μην τα λέτε λάθος. Εγώ είπα ότι θα πρέπει να είναι μια κατάσταση από την οποία βγαίνουν κερδισμένοι όλοι. Δεν είπα ότι βγαίνουν κερδισμένοι όλοι, γιατί προφανώς μας ανησυχούν οι πρόσφυγες τους οποίους επιστρέφουμε, τα άτομα τα οποία επιστρέφουμε και προσπάθησα στην προηγούμενη παρέμβασή μου να σας εξηγήσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επαγρυπνεί ούτω ώστε να ξαναδούμε τα όσα ισχύουν, τους κανόνες που ισχύουν στην Τουρκία σε ό,τι αφορά την υποδοχή των ε, προσφύγων στην Τουρκία. Είναι σκανδαλώδε αυτό το πινκ πον που παίζεται μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας για τους πρόσφυγες. Θα πρέπει απλώς να βελτιωθούν οι κανόνε υποδοχής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε. Και στη γραπτή ερώτηση αναφέρεται ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την οδηγία όχι τόσο επιθυμητή. Νομίζω ότι η συμφωνία είναι μια καλύτερη λύση. Ναι, Μία ερώτηση που δεν απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πόσα, πόσοι υπήκοοι τρίτων χωρών υπάρχουν. Τι γίνεται με την περίπτωση της Συρίας. Πόσα έχει διαδικασία έτσι. Αυτό δεν κατέστησε σαφές από την απάντησή σας. Παρακαλώ πολύ σύντομα κύριε Τουντοράτσε. Συμφωνείτε φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε να πούμε πόσες ε, ακριβώς επιχειρήσεις τέτοιες ε, και επιστροφής θα έχουμε. Ε, υπάρχουν ετούντες άσυλο που η αίτησή τους έχει απορριφθεί. Υπάρχουν περιπτώσεις που το κράτος μέλος αποφασίζει ποιος θα επιστραφεί και πού θα επιστραφεί. Είναι λοιπόν αδύνατον για μένα σε αυτό το στάδιο να σας πω ακριβώς κάποιο νούμερο πόσοι Τούρκοι υπήκοοι, πόσοι υπήκοοι τρίτων χωρών θα ε, έχουν επιπτώσεις από αυτό. Έπειτα, το θέμα είναι και πότε θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Εμείς θα ενημερώσουμε την Επιτροπή αυτή για το πότε θα γίνει και τότε θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες. Το σημείο όμως αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να σας πω κάτι ακριβέστερο. Κυρία Ζόμερ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία συνάδελφε, κυρία Ένστη, θέλω να σας πω ότι δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ακριβώς τα νούμερα, το πόσοι πλήττονται από αυτό. Κύριε Πρόεδρε, βλέπω πως όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν. Έχουμε έναν κοινό παρονομαστή. Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα δωράκι έτσι απλά στην Τουρκία. Και αυτό υπόθηκε. Αυτό θα ήταν όντως ανεύθυνο. Αυτό που επιθυμούμε είναι η Τουρκία να δείξει πως είναι ικανή να τηρήσει τις υποσχέσεις της, να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη. Και υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες ανησυχίες φυσικά για το ότι αυτοί οι πρόσφυγες, αυτοί οι μετανάστες θα σταλούν πίσω στην Τουρκία σε μια πολύ άσχημη κατάσταση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και όλα αυτά που έχουν ήδη υποθεί και όλα αυτά που φανταζόμαστε για το τι γίνεται εκεί πέρα. Η Συμφωνία Επανιστοχής όμως σε συνδυασμό με την ελευθέρωση των θεωρήσεων είναι κάτι το οποίο ε, είναι γεγονός και είναι κάτι το οποίο η Τουρκία στο τέλος θα αποφασίσει για το, για το τι θα γίνει, για το αν θα συνεχίσει γρήγορα, για το αν θα διακοπεί, για το αν θα υπάρξει παράταση, για το πώς θα συνεχιστεί αυτός ο διάλογος. Διότι σε τελική ανάλυση έτσι έχουν τα πράγματα και αυτή τη στιγμή ο διάλογος είναι το μόνο μέσο που έχουμε για να πιέσουμε την Τουρκία, για να τους πιέσουμε να ε, υπογράψουν και να εφαρμόσουν πλήρως αυτή τη συμφωνία επανιστοχής. Ε, και με αυτά τα λόγια θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επικοδομητική συζήτηση και ελπίζω αύριο να έχω μια στήριξη από εσάς έτσι ώστε να έχουμε ένα δυνατό ναι στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσία τους και τη συνεισφορά τους. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση του λίγου χρόνου που έχουμε. Θα συνεχίσουμε αύριο στις 9 το πρωί. Σας ευχαριστώ όλους. Γεια σας.